Bueno, buenas tardes. Ahora puerta. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με τη μερική διάταξη. Α περάσουμε στο σημείο 17, τροποποίηση του κανονισμού 1185 του 2003 σχετικά με την αφαίρεση των παιδιών καρχαρία επί των σκαφών. Στην τελευταία συνεδρίαση τη Επιτροπή, η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή τη και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την ε, γνωμοδότηση αυτή και χωρίς χρόνο τρεβή να δώσω το λόγο στην κυρία Πατράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή την πρώτη αντιλογή απόψεων. Επικεντρωνόμενοι σε δύο πτυχές που εγώ θεωρώ ως ε, προϋποθέσεις ε, τους σκέψεις μου. Καταρχήν να πω ότι αυτό το θέμα είναι συναισθηματικά φορτισμένο. Και φυσικά είναι και δικαιολογημένα αυτή η συναισθηματική φόρτιση. Αλλά πρέπει να το συνειδητοποιούμε αυτό το γεγονός και πρέπει και να συνειδητοποιούμε το ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ λανθασμένες και ελληματικές. Πολύ συχνά εγώ είδα ότι όταν μιλάω με ανθρώπους που θα έπρεπε να γνωρίζουν ε, το θέμα για το οποίο μιλάνε, δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα τι διακυβεύεται. Αυτή είναι μια πρώτη πτυχή που εγώ θα ήθελα να τονίσω εδώ δηλαδή στο ότι υπάρχει αυτή η συναισθηματικότητα και ότι υπάρχουν ε, πολύ ελληματικές πληροφορίες και λανθασμένες γιατί είναι σημαντικό να υπερβούμε αυτές τις δύο πτυχές προκειμένου η συζήτηση να μπορεί να γίνει σε ένα λογικό επίπεδο και αντικειμενικότητα. Τώρα, δεύτερη προπόθεση που θα ήθελα εγώ τώρα να αποσαφηνίσω εδώ είναι ότι από τη δική μου πλευρά σε σχέση με το θέμα αυτό, ακολουθώ μια μεθοδολογία όπως ε, συνήθως, δηλαδή να ακούσω όλα τα μέρη, να μελετήσω τα ζητήματα και να εντοπίσω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα που διακυδεύεται εδώ. Γιατί δεν είναι πάντοτε προφανές, κυρίως όταν οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς διακυβεύεται, ποιο είναι το ακριβές πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα δώσουμε μια λογική απάντηση που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των διάφορων ε, ενδιαφερομένων μερών και θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητο, απαραίτητα οι πιο απλές αυτές. Δηλαδή, Πολλές φορές ε, ο πιο απλός ε, και ο πιο γρήγορος δρόμος δεν είναι ο πλέον κατάλληλος ή ο πιο υπεύθυνο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι υπεύθυνο είναι να βρούμε μία λογική λύση για τα διάφορα συμφέροντα. Και βάσει αυτών των δύο προϋποθέσεων, αφού σας τις εγώ θα άρχισα να σας πω τι είναι αυτό το φίνινγκ, η αφαίρεση των πτεριγίων. Γιατί δεν μιλάμε για την αλίευση του καρχαρία όταν μιλάμε για φίνινγκ. Ε, την ε, κοπή των πτυριγίων ε, και για το ότι το σώμα του καρχαρία πετάγεται εκτός του σκάφους να είναι κάτι, ένα παρεμπίπτον αλίευμα. Αυτή είναι η πρακτική του φίνινγκ και έλαβα πολλά μέλη που έλεγαν ότι η πρακτική του φίνινγκ, δηλαδή τη αφαίρεση στο πτερυγείο, ήταν ακριβώ αυτό. Αλλά, ε, κοιτάξτε, η πρακτική του φίνινγκ είναι ότι εκμεταλλεύεται κάποιο τα πτερυγεία και κατόπιν πετάει το υπόλοιπο ζώο. Η πρακτική αυτή της αφαίρεση λοιπόν των πτερυγίων του φίνιγκ είναι απαράδεκτη από πολλαπλή σκοπιά, δηλαδή από περιβαλλοντική σκοπιά, ε, γιατί ουσιαστικά απειλεί ορισμένα είδη καρχαριών και είναι απαράδεκτη από κοινωνική και οικονομική σκοπιά, γιατί πραγματικά χάνεται ένα τρόφιμο με εμπορική αξία και από ηθική ε, σκοπιά είναι απαράδεκτο γιατί αποτελεί ε, μια πράξη που δεν σέβεται καθόλου ε, την ζωή του ζώου. Πρόκειται λοιπόν για μια παράδεκτη πρακτική. Όμω ε, είναι απαγορευμένη αφαίρεση των τεργείων, αυτό το φίνινγκ είναι απαγορευμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2003. Και ε, με συγχωρήσουν ε, όσοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα εκ των σύνεγγυς, όμως η αλήθεια είναι ότι από διάφορες ε, επαφές φαίνεται ότι υπάρχουν εδώ πολλές παρεξηγήσεις. Το φίνινγκ είναι απαράδεκτο και έχει απαγορευτεί από το 2003 και το 2005 το 2006 έχουμε έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Κοινοβούλιο που μας επιβεβαίωνουν ότι πράγματι δεν υπάρχει φίνινγκ στον ευρωπαϊκό τόλο. Τώρα, τι διακυβεύεται εδώ. Αυτό που διακυβεύεται με αυτή την πρόταση που λάβουμε από την Κομισιόν είναι να εξελιχθεί μια, παρά, μια ε, εξαίρεση. Όμως δεν είναι εξαίρεση το φίνικ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αποτελεί μια εξαίρεση το να κόβονται επί του σκάφους τα πτερήγια. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε. Τώρα, ποιε είναι οι επιχειρήσει οι οποίε χρησιμοποιούν αυτή την παρέκκληση. Είναι ο στόλος, ε, τα πλοία με κατάψυξη. Δηλαδή, εμεί έχουμε ένα στόλο που αλλιεύει κυρίως ε, δύο είδη και έχουμε το ένα είδος που αποτελεί το 80-90% ε, ε, είναι το απόθεμα αυτό υγιές, δεν έχει πρόβλημα και θα αλλιεύσει αυτά τα δύο είδη ο στόλος μας ε, και έχουμε ένα στόλο που μένει στη θάλασσα για ένα μήνα περίπου ε, και επομένως εφόσον παραμένει στη θάλασσα για ένα μήνα περίπου δεν ε, βάζει στην την κατάψυξη το ψάρι και επειδή δεν το βάζει στην κατάψυξη δεν χρειάζεται να ε, αφαιρέσει τα πτερίγια. Τώρα πότε γίνεται αυτή η αφαίρεση των πτερυγίων. Γίνεται αυτή η αφαίρεση των πτερυγίων από το στόλο που βάζει στην κατάψυξη το ψάρι, αυτή που παραμένει στη θάλασσα πάνω από ένα μήνα, περίπου τρει μήνε και η πρακτική αυτή της κοπής γίνεται από ένα μειονεκτικό κομμάτι του στόλου, μειοψηφικό με συγχωρείτε κομμάτι του στόλου. Δηλαδή αυτός ο στόλος ε, ε, προβαίνει στην κοπή των πτερυγίων για να αποθηκεύσει ξεχωριστά τα πτερύγια από το σώμα του ζώου. Ε, Γι' αυτό αυτός ο τομέας ε, θεωρεί ότι ε, η αφαίρεση των πτεργίων επί του σκάφους είναι κάτι απαραίτητο. Τα επιχειρήματα που αναφέρονται εδώ και εγώ θα πω τώρα ποια είναι τα πιο σχετικά, έχουν να κάνουν με την ε, ποιότητα του τροφίμου και την υγεία. Αν ε, καταψύχεται το ζώο επί του σκάφους. Χωρίς τα πτερίγια, όταν φτάνει στους ε, λιμένες, ε, τότε μπορεί να εκφορτωθεί από τη μία το σώμα, από την άλλη τα πτερίγια, μπορούν να εκφορτωθούν ε, και ακολουθούνται διαφορετικές εμπορικές οδοί και έτσι λοιπόν και τα δύο πρέπει να είναι καταψυγμένα μετά την αλίευση. Με αυτή την κατάργηση της παρέκκλησης εμείς θα είχαμε την εξής κατάσταση. Το ζώο θα καταψύχεται μαζί με τα πτερήγια μία από τις προτάσεις ε, της Επιτροπής είναι τα ε, να κοπούν με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να διπλωθούν πάνω ε, στο ε, σώμα όταν όμως ε, θα εκφορτωθεί στην ξηρά θα πρέπει να υπάρξει μερική απόψυξη του ζώου προκειμένου το πτερίγιο να μπορεί να κοπεί μέχρι το τέλος. Και όπως είπα πριν να διοχετευτεί σε άλλες αγορές. Τώρα αυτή η μερική απόψυξη όπως γνωρίζετε θα έχει επίπτωση έτος. Και θα σημαίνει ότι θα υπάρχει μείωση της τιμής της πώληση ε, του κρέατος του ζώου και φυσικά υπάρχουν και κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέμα που τονίζεται είναι το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή ότι τα καταψυγμένα πτερήγια λειτουργούν ε, ως... Ε, presas ao tronco do animal eh, implica Λειτουργούν λεπίδες και ε, έτσι λοιπόν ε, αυτό μπορεί να σημαίνει ε, κίνδυνο για την ασφάλεια του πληρώματος. Μιλάμε για ένα πλήρωμα σε ένα σκάφος το οποίο δεν είναι αραγμένο και υπάρχει μια δυσκολία στο χειρισμό του ζώου. Όταν τα πτερήγια μπορούν ε, να είναι αρκετά κοφτερά. Το ότι διπλώνεται το πτερίγιο και διπλώνεται όπως σας είπα πάνω στο σώμα, ελαχιστοποιεί αυτό ε, το πρόβλημα αλλά δεν το εξαλείφει όπως επίση ε, και το τύλιγμα σε πλαστικό και κάτι που δεν το κάνει ο συστόλος γιατί ε, δεν εξελίχθηκε το πρόβλημα γιατί έπρεπε να δούμε τι είδου υλικό χρησιμοποιείται για να μην ε, κόβεται και το υλικό αυτό. Έχουμε λοιπόν το θέμα της υγείας, το θέμα της ασφάλειας και δεν μπορώ παρά να αναφέρω και το θέμα της ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί αν ε, δεν υπήρχαν οι μεταποίησεις από τους σκάφους του ζώου, τότε θα διατηρούνταν τα ε, πτερίγια επί του σώματος και θα υπήρχε μεγαλύτερος χώρος από όσο χρειάζεται επί του σκάφους και αυτό θα σημαίνει λιγότερη βελτιστοποίηση του χώρου επί του σκάφους. Και αυτό θα αιτιολογούσε πιο συχνές ε, ε, μετακινήσει στους λιμένες προκειμένου να γίνει εκφόρτωση. Λοιπόν, τώρα, εμείς ερωτηθήκαμε γιατί παρουσίασε την πρόταση αυτή η Κομισιόν. Ο πρώτος λόγος που επικαλέστηκε η Κομισιόν και μπορώ να σας πω ότι εμένα με εξέπληξαν οι όροι με τους οποίους αναφέρθηκε, παράθεση είναι να εξαλειφθεί η ε, πρακτική, αυτή η τρομερή πρακτική ε, του να κόβονται τα πτερία και να ε, προστατεύονται καλύτερα τα ζώα. Δηλαδή να εξελίψουμε αυτή την τρομερή πρακτική της κοπής των πτερυγίων είπε η Επίτροπος. Και εδώ φαίνεται ότι είναι απαράδεκτη αυτή η πρακτική του φίνινγκ. Το μπερδεύουμε όμως αυτό με τη διαδικασία της αφαίρεσης των πτεριγίων αλλά εκμεταλλευόμενοι το σώμα του ζώου. Έτσι λοιπόν, τι, περιμέ, τι θέλει η Κομισιόν να πετύχει, να εξαλείψει το feeling. Όμως, Ε, η Κομισιόν ε, ε, έχει πληροφορίες για το feeling και η ΚΑΠΑΟ μας είπαν όχι, ότι δεν υπάρχουν ε, δεδομένα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να εξαλειφθεί αυτό το θέμα πρέπει να σκεφτούμε βάσει ποιων αρχών εμείς θέλουμε να λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις. Γιατί αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ε, και εμεί λαμβάνουμε νομοθετικές αποφάσεις, αυτό αντίκειται σε αυτό που λέμε εδώ, ότι χρειαζόμαστε να έχουμε όλο και περισσότερες τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες για να μπορέσουμε να λαμβάνουμε τις κατάλληλες ε, νομοθετικές αποφάσεις. Και ακόμη πιο ανησυχητικό είναι όταν εμείς ε, είμαστε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή ελευτικής πολιτικής και πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι αρχές που θα εφαρμόσουμε για αυτή τη μεταρρύθμιση που θεωρούμε ότι είναι σοβαρή και εις βάθος. Άλλα στοιχεία που αναφέρονται από την Κομισιόν, καλύτερη συλλογή δεδομένων και μία καλύτερη διαχείριση των αλλιευμάτων. ενώπιον ε, των πτυχών αυτών. Και φυσικά ε, δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα σε αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ούτε τα επιχειρήματα, ούτε τις ε, πληροφορίες και ελπίζω να εργαστώ με όλους τους κοιόδες συζητητές προκειμένου να βρούμε μέτρα πιο κατάλληλα και που δεν θα είναι απαραίτητο και τα πλέον απλά Όπω σα είπα, είχαμε και επαφέ με ένα μεγάλο μέρο ε, των σχεδόν συγητών για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ε, στην εξέβρεση πιο κατάλληλων λύσεων. σε αυτού λοιπόν. Ε, να πω ότι αυτή η κατάργηση της παρέκκλησης που προτείνεται τώρα από την Επίτροπο προκαλεί μια πραγματική ζημία στο στόλο των πλοίων με κατάψυξη. Και είναι ακριβώς αυτός ο στόλος που χρειάζεται αυτή την παρέκκληση. Και πρέπει να υπάρχει επαρκής νομοθεσία για να υπάρχει έλεγχος υγειονομικός. Και είναι κάτι θεμελιώδες εδώ αυτό. Τώρα, κατόπιν ε, αυτής της ε, σύντομης έκθεσης ιδεών, θα ήθελα εδώ να προτείνω καταρχήν. Εξή. Καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια δεδομένα για την ύπαρξη του φίνινγκ και καθώ η πρόταση αυτή τη Κομισιόν δεν είναι κατά του φίνινγκ γιατί έχει ήδη απαγορευτεί αλλά είναι κατά μια υποψία ύπαρξη φίνινγκ Λοιπόν, γνωρίζοντα ότι υπάρχουν πραγματικέ ζημίε για το στόλο, γνωρίζοντα επίση ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία ε, σε ένα στάδιο μεταρρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική και όλοι ξέρουμε ότι οποιοδήποτε και αν είναι ο προσανατολισμό που θα ακολουθηθεί, θα έχουμε πολύ βαθιέ μεταρρυθμίσει, πολύ βαθιέ αλλαγέ στον τομέα τη αλληλεία και αυτό θα σημαίνει λιγότερα σκάφη και λιγότερου αλληλεί, γιατί Ζούμε τώρα σε μια κατάσταση πραγματικής πίεσης που ασκείται στον ληφτικό τομέα, στον ληφτικό κλάδο. Να ρωτήσω, ε, μήπως θα έπρεπε να διατηρήσουμε την παρέκκληση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταρρύθμισης της ε, πολιτική, πολιτικής, έτσι ώστε να μην αυξήσουμε περισσότερο την πίεση στον κλάδο που αυτή τη στιγμή πραγματικά βιώνει μια διαδικασία μεταρρύθμισης ε, και αναδιάρθρωσης για να μπορέσει να επιβιώσει στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης, να μην ε, προσθέσουμε ένα ακόμη επιβαρυτικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα να διατηρήσουμε την παρέκκληση. Μέχρι να εφαρμοστεί η κοινή ελευτική πολιτική προκειμένου να μην δημιουργήσουμε έναν ακόμη παράγοντα άσκησης πίεσης, συμφόρησης στον τομέα και για να μπορέσουμε να καταστήσουμε δυνατή την απόκτηση των δεδομένων αυτών που όλοι λένε ότι δεν έχουμε και θα ήταν πιθανό ότι αν τα είχαμε θα μπορούσαμε να λάβουμε και μια πιο κατάλληλη θέση. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μία συζήτηση και για άλλα μέτρα που να αφαιρούν το βάρος της απόδειξης ε, για το Φίνινγκ από τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Και ορισμένες ιδέες για μελλοντική συζήτηση θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από την εξέλιξη των ειδικών αδειών αλίας. Αναφέρατε αυτό στην παρέκκληση για το στόλο που αλεύει νοπά ψάρια. ή το να γίνουν παραδεκτές αυτές οι ειδικέ άδειε ελίας μόνο για τα πλοία κατάψυξη, αλλά αυτά που εφαρμόζουν, αυτοί που εφαρμόζουν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας που μας επιτρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ότι τα πτερίγια ε, έχουν αφαιρεθεί από κάποια σώματα καρχαρία τα οποία και αυτά εκφορτώνονται. Και μάλιστα σε αυτό τοποθετήθηκε σχετικά και η Άλλη πτυχή που θα μπορούσε να συζητηθεί είναι ο υποχρεωτικό χαρακτήρα τη ταυτόχρονη εκφόρτωση των πτεργείων και των σωμάτων των καρχαριών ω ένα τρόπο ενίσχυση του ελέγχου. Γιατί εμείς ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τον έλεγχο για να είμαστε σίγουροι ότι θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η υποψία. Άλλη πτυχή. υποχρεωτικό χαρακτήρας ε, εκμετάλλευση όλων των μερών του Καρχαρία και τη ουράς ε, και όλου του σώματος και δημιουργία σχεδίων διαχείρισης και αλίευσης για να απαντήσουμε στις ανησυχίες της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ελευμάτων. Ακόμη και αν εμείς γνωρίζουμε το 80-90% όπως σας είπα ε, Μπριονάς ε, γκλάουκα στα λατινικά, είναι αυτό το είδο. Και μια άλλη ιδέα που θέλω να αναφέρω εδώ είναι η εφαρμογή σε όλες τις ε, περιφερειακές οργανώσεις αλίας ενός προγράμματος στατιστικής τεκμηρίωσης για την εμπορία των πτερυγίων καρχαρία. Και εδώ για μια ακόμη φορά να πω ότι η συζήτηση αυτή έγινε και στην ΕΟΚΕ. Λοιπόν, είχατε πολύ μεγάλη υπομονή μαζί μου, Πρόεδρε, να κλείσω εδώ. Να πω ότι πέρα από την αρχική πρόταση, αυτές οι πτυχές που παρουσιάζω εδώ για να συζητηθούν έχουν ως στόχο όχι να συμμορφωθούμε με τις πιο απλές λύσεις, αλλά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή να ακούσουμε τον τομέα, να ακούσουμε τον κλάδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πιο κατάλληλες λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πατρά. Κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Πατράου Νέβες ε, για τις αγωγικές παρατηρήσεις ε, που έκανα. Ε, είχαμε μία σύσκεψη χτες το βράδυ με την κυρία Πατράου Νέβες γιατί είμαι σκιώδης για την πολιτική μου ομάδα για το θέμα αυτό και θέλω ολόκληρα να την ευχαριστήσω διότι ε, ακολουθεί, προσεγγίζει συλλογικά το θέμα, πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία γιατί είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα το ζήτημα και κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να έρθει σε τακτική επαφή με όλους τους κοιόδης. Επίσης χαίρομαι διότι ε, με πυγμή υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας σας γιατί κυρίως Πορτογαλία και Ισπανία είναι που αλλιεύουν καρχαρίες και καρχαροειδή. Ε, είμαστε από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς και πτερυγίων και κρέατος με ηγέτες ε, φυσικά την Ισπανία και την Πορτογαλία ως προς τον όγκο εξαγωγών και δεν με ξαφνιάζει ε, που προτάσει την ασπίδα της και υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα για να μην περάσει για να κλείσουμε αυτό το παραθυράκι που αφήνει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. το βράδυ μου έλεγε η κυρία Πατράου ότι η εξαίρεση που έχουμε εφαρμόσει ούτω ώστε να επιτραπεί η αφαίρεση εν πλώ των ε, πτερυγίων χρησιμοποιείται μόνο από ελάχιστο ε, αμεληταίο αριθμό σκαφών ε, ε, δηλαδή σκάφη με καταψύχτες που μένουν στη θάλασσα τρεις μήνες ε, συγκεκριμένα και αν επιμείνουμε να εκφορτωθεί ολόκληρος ο Καρχαρίας με άθικτα τα πτερήγια του θα έχουμε σοβαρά προβλήματα όπως μας έλεγε προηγουμένως. Εγώ πίεσα την κυρία Πατράου όταν ε, ε, είπαμε ότι προ... μιλάμε για λιγότερο από 20 σκάφη. Κοιτάξτε, όταν πήγα τελευταία φορά στο Βίγκο είδα δύο πυραμίδες ε, από μπλε καρχαρίες που εκφορτώθηκαν με τα πτερίγια τους και αυτό καταδεικνύει, μου είπε, ότι η εξαίρεση είναι απαραίτητη αποκλειστικά και μόνο για αμεληταίο αριθμό σκαφών και σίγουρα δεν εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αλίευσης καρχαριών και καρχαριοειδών. Αντιλαμβάνομαι τώρα από αυτό που μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία υπέβαλαν αίτηση για 200, 200 εξαιρέσεις, 200 άδειε δηλαδή για σκάφη Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητούμε γίνεται, υποβάλλονται αυτές οι αιτήσει. Ε, καταλαβαίνετε ανάμεσα στο 20 και τα, τα 20 σκάφη και τα 200 είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα. Θέλω να ξέρω τι συμβαίνει λοιπόν. Εάν δεν υπάρχει ε, τεκμηρίωση παράνομης δραστηριότητας και αφαίρεσης επτεριγίων εν πλώ, ε, ας με ενημερώσετε. Αλλά όσο υπάρχει αυτό το παραθυράκι θα υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα παράνομης αλίας ειδών, διότι Πρέπει να καταλάβετε πως γι' αυτό το λόγο ανησυχούν πολύ. Θέλουν να ε, κλείσουν αυτή, αυτό το παραθυράκι. Εγώ χρειάζομαι πολύ ε, κρατεότερες αποδείξεις. Όχι να μου πείτε ότι υπάρχουν 20-25 ε, πλοία καταψύχτες που θα χρειαστούν την εξαίρεση και προτού εγώ αρχίσω λίγο να το βλέπω πιο άνετα το θέμα, να σοκάρομαι και να μαθαίνω ότι υποβάλλανε αίτηση για 200 άδειε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού, ενεργειακής απόδοσης, θέμα επανάψυξης του καρχαρίου, Όλα αυτά που αναφέρατε είναι, είναι ουσιαστικά ζητήματα. Έχω δει σε πολλά ρεπορτάζ, ε, ε, εκπομπές ε, της τηλεόρασης. Στην Ασία εκατοντάδες καρχαρίες στην παραλία να στεγνώνουν στον ήλιο, οπότε ε, ε, η απόψυξη, η αφαίρεση πτερυγίων και επανάψυξη όταν μου λέτε ότι δημιουργεί πρόβλημα υγειονομικό δυσκολεύομαι να το φανταστώ σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου τέλος πάντων θα παραμείνω ανοιχτό σε περαιτέρω συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε. Αλλά σίγουρα ανησύχησα μόλις άκουσα αυτούς τους αριθμούς. Ο κύριος Δρομέο. Eh, η κυρία Πατραονέβες ξεκίνησε λέγοντας ότι αυτό είναι ένα θέμα φορτισμένο συναισθηματικά και μας ζήτησε να κάνουμε μία ανάλυση βασισμένη σε γεγονότα. Εγώ αυτό θα προσπαθήσω να κάνω βασικά, γιατί το πρόβλημα, του ουσιαστικό για μένα, είναι ότι το πρόβλημα είναι απλό. Η λύση που υπάρχει σήμερα είναι πολύπλοκη και φοβάμαι ότι η λύση τη χειρής πατρονεύης είναι ακόμη πιο πολύπλοκη. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Ας ε, ξεκινήσουμε από τη βάση ότι οι καρχαρίες ε, και τα λεσμοβράχια ήδη, τα σελάχια, οι καρχαρίε κτλ. είναι πολύ ευπαθή, ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της διάστασής τους ε, σε βιολογικό επίπεδο, λόγω των χαρακτηριστικών τους. Δηλαδή, τι γίνεται τελικά, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το είδους πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ να, τη στιγμή που θεσπίζουμε τα μέτρα διαχείρισης ε, για αυτά τα αλίευματα. Δηλαδή, όχι μόνο να του επιτρέψουν να φτάσουν ε, σε ορίμανση για να αναπαραχθούν, αλλά ε, υπάρχουν ε, δύο παραδείγματα. έχουμε. Παραδείγματος χάρη αυτό το γραφικό καρχαρία που αναφέρατε. Που είναι το είδος που αλλιεύεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η UCN θεωρεί ως ένα ευπαθές είδος, ένα ευάλωτο είδος στη Μεσόγειο και απειλείται ε, στον κόσμο και έχουμε και ένα άλλο είδος ε, καρχαρία ε, το οποίο επίσης θεωρείται ευάλωτο. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Εδώ σε κάποιο βαθμό πρέπει ε, να διευκολύνουμε ένα τμήμα του στόλου. Είδαμε ότι αυτό αφορά κυρίως τα πλοία καταψύκτες και όχι τα πλοία που αλεύουν οπά. Το άλλο είδε στον Καρχαρίας Λάμνα. Ε, μιλάμε και για θέματα ηθικής. Όταν ε, έχουμε ένα σύστημα που ότι ορισμένες χώρες ε, εφαρμόζουν, το χάρη, το 5% της αναλογίας του βάρους ε, σε σχέση με το ζωντανό βάρος και άλλοι χρησιμοποιούν το 5% του καθαρού βάρους, έχουμε ένα πρόβλημα και υπάρχουν αποκλήσεις. Το δεύτερο πρόβλημα είναι πώς το υπολογίζουμε αυτό. Ήδη από την αρχή είναι δύσκολο, είναι πολύπλοκο για να μην πούμε ότι είναι αδύνατο. Η πρόταση της κυρίας Πατραονέβες είναι ότι θα τα καταστήσουμε πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Επομένως εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε αυτήν την κατεύθυνση ότι δεν είναι κάτι σωστό. Λοιπόν, τρίτο τώρα σχόλιο. Αν το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι το σημερινό σύστημα δεν μας ε, εγγυάται ένα λογικό σύστημα διαχείρισης ε, που να συνάδει με το στόχο του να διατηρήσουμε τα τα επίπεδα ε, των ζώων σε ο επιθυμητό, για μένα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τελικά να εθετήσουμε την πρόταση γιατί μα ε, οδηγεί σε αυτό που ζήτησε η κυρία Πατρεωνέβες, δηλαδή στι πληροφορίε. Γιατί αν ξεχωριστά εκφορτώνουμε το σφάγιο από τα πτερίγια έχουμε πρόβλημα λογιστική και θα έχουμε πρόβλημα να ξέρουμε για ποια είδη μιλάμε, για πόσα ζώα έχουμε και στην πραγματικότητα ποιε είναι οι διαστάσεις αυτού του ελιεύματος. Αν ε, έχουμε τα πτερίγια μαζί στην εκφόρτωση δεν έχουμε ε, το ίδιο πρόβλημα. Δεύτερον, αναφέρθηκαν ορισμένε συγκεκριμένε στοιχείε όπω η ασφάλεια. Αυτό είναι λυμένο λύνεται. Αν τα πτερίγια διπλώνονται και δένονται πάνω στο σώμα, δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας μέσα στο σκάφος. Τρίτο πρόβλημα. Το θέμα το υγειονομικό τη υγιεινή. Αν δεν κάνω λάθο και αν έχω σωστέ πληροφορίε, πιστεύω πω ναι, και αυτό το πρόβλημα λύνεται γιατί μπορούμε να κόψουμε ως ένα σημείο το πτερίγιο και αυτό επιτρέπει με φυσικό τρόπο το πτερίγιο να κολληθεί πάνω στο σώμα που αυτό ζητάμε και όταν έχει καταψυχθεί να το κόψουμε πλήρως το πτερίγιο, αυτό είναι δυνατό, έτσι λοιπόν δεν σπάει και η λυσίδα του ψύχους και είναι δυνατό να γίνει αυτό, έχει αποδειχθεί ότι είναι εύκολο να γίνει και έτσι δεν έχουμε αλλίωση της Αλυσίδα του ψύχους. Και το κάνουν ορισμένες χώρε και εμείς ε, θα είμαστε εξαίρεση αν δεν το κάναμε. Τέταρτη και τελευταία σκέψη προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν το ανέφερε η κυρία Πατρέων Εύες, αλλά αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που επίση ε, τίθεται συνήθω το ότι έχουμε στόλου που είναι στη θάλασσα για πολύ καιρό και έτσι είναι δύσκολο να διαχειριστούν δύο προϊόντα που έχουν διαφορετικές αγορές, δηλαδή ε, το σώμα του καρχαρία, το σφάγιο και τα πτερίγια. Ε, αυτό το θέμα επίσης λύνεται τόσο με το χειρισμό, ε, με την εκφόρτωση ολόκληρου του σώματος ε, σε ένα ε, λιμένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το πιστοποιητικό προέλευση στο ευρωπαϊκό. Αυτό μπορεί να διατηρηθεί, δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Επίσης, από τη σκοπιά της πρόσβασης σε άλλες αγορές μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις σε άλλες αγορές. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Από την οικονομική σκοπιά Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει κάποια δυσκολία για τον κλάδο, όμως θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε με ακρίβεια ποιο είναι ο υποτιθέμενο οικονομικό κίνδυνο, ποιε είναι οι συγκεκριμένε οικονομικέ ζημίε που θα επαληθούν. Εγώ δεν είδα κανένα νούμερο στην κατεύθυνση αυτή, αριθμητικό στοιχείο. Και είπε και η κυρία Πατρεωνέβα ότι γενικά θα χαθούν θέσει εργασία, ε, αλλά θα μειωθούν και τα σκάφη. Θα ήθελα όμω μία εκτίμηση οικονομική. Δεν την είδα, δεν νομίζω να είναι και τόσο μεγάλη αυτή η απώλεια, αυτή η ζημία και από τεχνική σκοπιά όλα τα προβλήματα που τέθηκαν έχουν επιληθεί. Συμπέρασμα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω καμία λύση παρά να υποστηρίξουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της Κομισιόν που απλώς ε, καθιστά πιο εύκολη πιο εύκολο και πιο συνεκτικό τον χειρισμό τέτοιου είδους αλλιευμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Ρωτάει ο εισηγητής ε, γιατί παρόλα αυτά προχωράει με την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, ε, Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει όταν πριν από 5-7 χρόνια κατέθεσαν την αρχική πρόταση. Του το είπαμε ότι θα έχει προβλήματα Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε, σα τα λέγαμε εμεί ε, τώρα που προέκυψαν τα προβλήματα. Λοιπόν, ας πάρουμε την αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, νομίζω εκεί βρίσκουμε πολλές απαντήσεις για όλες αυτές τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Όπως ξέρουμε, ο αρχικός ε, κανονισμός που κάποιοι από μεταξύ μου ε, επέκριναν ε, αναφέρει ότι μπορούν να εκφορτωθούν σε ξεχωριστούς λιμένες τα πτερίγια και ο κορμός. Ε, όχι ότι απαραίτητα πρέπει να προσδιοριστούν εκ των προτέρων τα λιμάνια, μπορεί και να μην έχει επιθεωρητές μπορεί και εμένα να έχει προβλεφθεί. Αυτό τέλο πάντων στον κανονισμό δεν υπάρχει καμία αμνία για παρουσία επιθεωρητών. Λέει επίση η έκθεση ότι είναι αδύνατο να τεκμηριώσουμε ότι δεν έχει προκύψει αφαίρεση πτερυγίων και πρέπει να βασιστούν ε, αυτοί που θα αποφανθούν αποκλειστικά και μόνο στο ημερολόγιο του πλοίου. Συγγνώμη, αλλά παραποιούνται τα στοιχεία. Τι κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλή μα. Όλοι, όλοι, όχι μόνο Πορτογαλική, Ισπανοί και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, την περασμένη εβδομάδα 17 σκήπε ε, κατηγορήθηκαν για μαζική απάντη υπεραλίευση. 16 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια ευρώ σκουμπρί και είναι τεράστια απάτη. Ε, παραποίηση στοιχείων, ε, οι πλάστικες, τι ηχθιόσκαλε, ό,τι θέλετε τέλο πάντων, μαζική απάτη. Ε, δηλαδή, το λέω αυτό για να μην, ε, να μην θεωρήσετε ότι κατηγορώ τους άλλους και όχι τη χώρα μου. Είμαστε εξίσου ένοχοι. Λοιπόν, στην έκθεση αξιολόγου λέμε Πέντε κράτη-μέλη έχουν αναφέρει διάφορες περιπτώσεις παραβίασης του κανονισμού. Γι' αυτό λοιπόν κατέθεσε προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα του καρχαριού αν είναι απειλούμενο είδος και τα λοιπά, για κάποιους ως όχι. Για τους ε, ρίγχο καρχαρίες δεν νομίζω να ε, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι απειλούμενο είδος. Δεν έχουμε επαρκή επιστημονικά στοιχεία ούτως ή άλλως. Όταν μιλάμε για τους γλαύκο καρχαρίες, τα λέω καλά, ε, για αυτούς τους καρχαρίες υπάρχει ανησυχία για την ε, διατήρηση του αποθέματος, αλλά τόσο πάνω κρεμεί το, το ζήτημα και συνεχίζονται τις συζητήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα. αντί να έχουμε ξεχωριστά τα πτερίγια και το σώμα του καρχαρία, Λέτε εσείς, λέει η συγκήτρια ότι πρέπει να τεμαχίσουμε, ε, αλλά όχι 100% του πτερίγιου το και να το διπλώσουμε. Υπάρχουν πρακτικές λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κύριε Ρομέντα ε, θα σας έλεγα ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν έχουν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με επιπρόσθετο κόστος που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η αλληλεία ε, του Ισπανικού και Πορτογολικού στόλου. Ούτε έχει τεκμηριωθεί αρνητική επίπτωση για την απασχόληση λόγω της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό. Η Κωνσταντίνα το κάνει, ναι. Ε, και σας ξαναλέω ότι λύσεις υπάρχουν για τα προβλήματα γιατί δεν περνάμε κατευθείαν στι λύσει και το συζητάμε κυρία Φράγα. Λοιπόν, και εγώ θέλω να είμαστε κάπως πιο ψυχρεμοί στο θέμα αυτό, γιατί εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να το δούμε στην δυνατόν πιο επεύθυνο και πιο λογικά. Αυτό το θέμα Κυρίω το κινούν μικρών περιβαλλοντικές και το γνωρίζουμε. Βέβαια είναι πλήρες δικαιωμάτους. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό, γιατί αν κάποιος διαβάσει όλες τις πληροφορίες που μας στέλνουν αυτές οι ΜΚΟ μικρών, πίσω από αυτές βρίσκεται η συνεχής υποψία ότι ο ευρωπαϊκό στόλο κάνει, προβαίνει σε φίνινγκ, δηλαδή ότι κόβει τα πτερίγια και πετάει τα σώματα των καρχαρίων στη θάλασσα. Και μάλιστα μέχρι και η Επίτροπος ε, το είπε, δεν χρειάζεται δηλαδή να δούμε την έκθεση των ΜΚΟ, ε, το είπε και η ίδια Επίτροπος. Εγώ πρέπει λοιπόν να πω ότι ε, για το καρχαρίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλο, όπως και το χείρο. Ε, δηλαδή από, ε, ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το έλαιο που χρησιμοποιούμε εμείς οι γυναίκες για τις ρητίδες και βγαίνει από τον Καρχαρία. Έτσι λοιπόν δεν πετάμε τίποτα, όλα όλα χρησιμοποιούνται όπως και χρησιμοποιούμε και το γουρούνι στο σύνολό του. Έτσι λοιπόν. Αν υπάρχει και, αν υπήρχε μόνο μία περίπτωση όπου μία μη όμικρον μπορούσε ε, να ε, πράγματι ότι γίνεται αυτό το Φίνινγκ θα το ξέρουμε. Κοιτάξτε, και δεν υπάρχει. Έχουμε τα παρασυρώμενα δίκτυα κάθε χρόνο. Έχουμε εκθέσεις με τους αριθμούς των σκαφών στη Μεσόγειο κτλ. Στην περίπτωση του φίνινγκ, ο κοινοτικό στόλος δεν έχει παρουσιάσει μία και μόνο περίπτωση κανένας ε, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αποδείξεις. Πρόκειται μόνο για υποψίες. Και αν μου πει κάποιος ποια είναι η ΚΟ που έχει μία απόδειξη. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για την πρακτική του φίνιγκ. Και δεν υπάρχει γιατί επιμένω ο κοινοτικό τόλος πολύ πριν από την ευρωπαϊκή ρύθμιση δεν ε, προέβαινε σε ε, γιατί θέλει να χρησιμοποιεί και τα πτερίγια αλλά και τον κορμό και το σώμα. Και τώρα σε ό,τι αφορά την ε, βιωσιμότητα, εγώ διάβασα την ε, έκθεση της ε, Οσεάνα και κοιτάξτε, αν κάποιος δεν ξέρει, οι καρχαρίε είναι 400 διαφορετικά είδη. Έχουμε κάποιους που είναι, κινδυνεύουν από εξαφάνιση, έχουμε άλλου καρχαρίες που είναι καρχαρίες βαθέων υδάτων κτλ. Και το κύριο είδος που είναι ο γλαυκοκαρχαρίας είναι ένα είδος ε, το οποίο αλλιεύεται στον Ατλαντικό και ε, στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ε, και όχι στη Μεσόγειο και βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Δηλαδή αυτό το λέει και το ΙΚΑΤ. Στόλος με με τα παραγάδια ε, ψαρεύει στους ωκεανούς. Και απαντάω τώρα στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος. Ο κύριος Στίβενσον. Υπάρχουν ε, ειδικέ αδείε για 41 ισπανικά και 10 πορτογαλικά σκάφη. Και ε, στόλος που είδατε εσείς ε, στο Βίγκο είναι τα παραδιαγδιάρικα που αλλιεύουν οπά ψάρια και πραγματικά από κοινού εκεί αυτοί εκφορτώνουν ε, και τα πτερίγια και τα σώματοκορχαρία δεν έχουν να κρύψουν τίποτα γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα αποθήκευσης όπως έχουμε στα πλοία κατά Έτσι λοιπόν το θέμα της βιωσιμότητας των ειδών αυτών, ε, κυρίως του κλευκοκαρχαρία, δεν υπάρχουν αυτό το αναγνωρίζει μόνο η Κομισιόν. Ε, τώρα η Ουσιάνα λέει ότι πρόκειται για ευάλωτα είδη και μιλάει γενικά. Όμω, ε, δεν ε, αναφέρει συγκεκριμένα είδη που αλλιεύει ο κόσμος τόλος. Έτσι λοιπόν μας οδηγεί η έκθεση αυτή σε πλάνη και σε μία παρερμηνία. Σε ό,τι φορά τώρα την αναλογία. Ναι, εγώ συμφωνώ. Ήδη υπήρχαν προβλήματα στην Νότια Αφρική. Και τα προβλήματα προέρχονται από την αναλογία. Γιατί η σύσταση του ICAT που ε, τη ζώνη εκεί λέει ότι ε, υπάρχει ένα ποσοστό 5% αλλά δεν διευκρινίζει αν είναι ζωντανό βάρος ή όχι και αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Μιλώ για τη σύσταση του ICAT και αυτό οδήγησε πολλές φορές ε, σε προβλήματα ερμηνείας. Δεν λέω εγώ λοιπόν ότι δεν πληρείται μερικές φορές η αναλογία, λέω... Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι ποτέ δεν έχει γίνει και το φίλινγκ, λέω ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις τέλος πάντων. Και αυτό που μα μπερδεύει περισσότερο είναι η σύσταση του ΙΚΑΤ, η οποία δεν προσδιορίζει αν πρόκειται για ζωντανό βάρο ή όχι. Η πρόταση ως έχει και κατόπιν ε, μπορούμε να περάσουμε στην ανάλυση του συμβασμού που προτείνει κυρία Πατράο. Η σημερινή πρόταση επιτρέπει την εκφόρτωση σε διάφορα λιμάνια, γιατί μιλάμε για διαφορετικές αγορές και μπορεί να έχουμε προβλήματα ελέγχου. Μπορώ να το κατανοήσω αυτό, ότι έτσι ως έχει μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, όμως η πρόταση της κυρίας Πατράο δεν είναι μια πρόταση που μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη, γιατί ζητείται καταρχήν μια παρέκκληση χρονική. Δηλαδή, μετά θα αναλυθεί εκ νέου το ζήτημα. Δεύτερον, δέχεται ότι ο στόλος ε, νοπών ε, ψαριών ε, μπορεί να εκφορτώνει μαζί πτερήγια και σώμα και για τους καταψύκτες, τα πλοία καταψύκτες ζητείται να μπορούν να εκφορτώνουν στον ίδιο λιμένα το σώμα αφενός και τα πτερήγια φετέρων και να υπάρχει ένα σύστημα ίχνηλασιμότητας που να είναι ένα ενδιάμεσο σύστημα μεταξύ αυτού που εφαρμόζει το ΕΚΑΤ και αυτού που εφαρμόζει η Κάμελαρ που είναι το πλέον ιδανικό. Έτσι λοιπόν με αυτό για μία περίοδο θα μπορούσαμε να έχουμε τις επαρκείς εγγύησεις προκειμένου να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λεχθέντως αυτού, συγγνώμη κυρία Ντέιβις, ε, θα στραφώ και πάλι σε εσά, αλλά εγώ διάβασα το είναι αξιολόγηση αντικτύπου και ακριβώς εκεί στο αξιολόγηση αντικτύπου η επιλογή που διάλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που κοστίζει πολύ για τα παραγαδιάρικα. Δεν θυμάμαι τώρα τα αριθμητικά στοιχεία και γι' αυτό δεν σας τα πω τώρα κύριε Ρουμέβα, αλλά λένε ότι πρόκειται για την πλέον δαπανηρή επιλογή που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, ως προς το κόστος. Λοιπόν, η κυρία Πατράου τα ξέρει καλύτερα από μένα. Ελπίζω ότι με αυτά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ένα συμβασμό που να Μα διευκολύνει. Ξέρουμε ότι μιλάμε για σπανικό και πορτοκαλικό στολό κύριε Στίβενσον, αλλά το θέμα είναι να διευκολύνουμε ε, αυτούς που σέβονται τους κανόνες. Ε, α, φυσικά αν ο γλαυκοκαρίας βρεθεί σε δίνει κατάσταση θα σταματήσουμε την αλίευση, θα σταματήσουμε στο τη αλίευση. Αλλά δεν υπάρχει τώρα τέτοιο θέμα βιωσιμότητας και τα προβλήματα του ελέγχου μπορούν να λυθούν με την πρόταση που μας έκανε η κυρία Πατράου εγώ ελπίζω να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό για το καλό όλων. Συμβιβασμού που να μας ικανοποιούν όλους και να μας δουν και εγγύσει για τους ελέγχους, γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν οι περισσότερες αμφιβολίες για τους καρχαρίες. Gracias, señora Fraga. Ο κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι νέος ε, βουλευτής, νέο μέλος της Επιτροπής και νέος βουλευτής στο Κοινοβούλιο. Πρώτη φορά έρχομαι σε συνεδρίαση και πρώτη φορά ζήτησα το λόγο. Και τον ζήτησα το λόγο για να ζητήσω συγγνώμη από πλευρά του Κρήτον Αρσένη, που είναι ο σκιώδη μα ε, για αυτό το θέμα. Δυστυχώ δεν μπορούσε να έρθει στη σημερινή συνεδρίαση. Έπρεπε να πάει και να παραμείνει στην Αθήνα διότι είναι και ο Μάρτιν Σούλτ σήμερα. Θα παρουσιάσω όμως εγώ την θέση του στο θέμα αυτό. Και θα το κάνω στα αγγλικά γιατί μου έδωσε τη σημειώση στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να καλωσορίσουμε θερμά τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διότι κλείνουν όλα τα παραθυράκια που υπήρχαν στον κανονισμό του 2003 και εξασφαλίζει ότι η αφαίρεση πτερυγίων δεν θα γίνεται πλέον εν πλώ σε σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εν πάση στα ύδατα της Ένωσης ε, μας ικανοποιεί η διαγραφή συγκεκριμένα του άρθρου 4 του κανονισμού 2003. Εκεί στο άρθρο 4 δινόταν η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χορηγήσουν ειδικέ αλληλευτικές άδειες που επιτρέπουν στα σκάφη να αποκλίνουν από την γενική απαγόρευση σχετικά με την αφαίρεση των πτερυγίων ε, εν Ε, όταν μιλάμε για ειδικέ ε, άδειε, επιτρέπεται η αφαίρεση των πτερυγίων, επιτρέπεται η εκφόρτωση και ε, σε διαφορετικέ χρονικέ τιμέ και σε διαφορετικά λιμάνια μπορούν να εκφορτώνονται αντίστοιχα τα πτερύγια και ο κορμό. Ε, σχεδόν αδύνατο ο έλεγχο, δηλαδή, γιατί η μόνη βάση για να κρίνουμε είναι τα ημερολόγια πλοίου. Έξω και τα παραθυράκια, έξω και οι παραβιάσει που σημειώθηκαν και λόγω των οποίων ε, η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών δεν επέτρεπαν πλέον ε, να ε, γίνει αφαίρεση εν πλώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ήταν μεταξύ των λίγων κρατών που χορήγησαν αυτές τις ειδικέ αλλιευτικέ άδειε. Διέκοψαν όμως αυτή την πρακτική τα τελευταία χρόνια λόγω θεμάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την υλοποίηση τη κείμενη νομοθεσία Επιπροσθέτω. Η έγκριση ε, της ε, μεθόδου για διάφορα είδη από διάφορα κράτη-μέλη και διάφορους διεθνείς οργανισμούς, ε, συγκεκριμένα και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Προστασίας των Καρχαριδών και 8 χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και η Ταϊβάν, σχάτως, απαγόρευσαν την αφαίρεση των πτερυγίων εν πλώ και τελικά αποφασίστηκε να παραμένουν τα πτερύγια. Ε, χρησιμοποιείται και ένας ε, λόγος, δηλαδή το ειδικό βάρος των πτερυγίων σε σχέση με το βάρος ολόκληρου του σώματος. Υτίθεται και το ζήτημα του υπολογισμού αυτού του αριθμητικού ε, λόγου που ούτως ή άλλως είναι διπλάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στον Καναδά και σε άλλες ε, χώρες Οι αλείς έχουν ε, ε, δικαίωμα να αλλιεύουν δύο με τρεις ε, καρχαρίες για κάθε έναν που εκφορτώνεται και καλούνται να μην υπερβαίνουν αυτόν τον λόγο του βάρους των πτερυγίων επί του βάρους των, του κορμού των καρχαρίων. Η ICC-AT παρεμποδίζει την εξέβρεση παγκόσμιας λύσης για αυτό το θέμα Ε, επίσης, ε, ε, αυτός ο διεθνής οργανισμός αναφέρει ότι δεν τηρούνται τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με το βάρος των καρχαριών που επιτρέπεται να εκφορτωθούν και μας καλούν να δώσουμε το παράδειγμα και όχι να έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα. Σε σχέση τώρα με τον κανονισμό του 2003 προβλέπονταν και οι υποχρεώσεις ε, υποβολής αναφορών δεν συμμορφώθηκαν όλα τα κράτη-μέλη και έχουν καταγγελθεί ε, περιπτώσεις. Το παράρτημα 3 της αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 αναφέρονται αυτές οι παραβιάσεις και σχετίζονται με αφαίρεση των ε, πτερυγίων και άρα παραβιάζεται η ευρωπαϊκή απαγόρευση αφαίρεσης ε, των πτερυγίων. Ο απότερος στόχος ε, είναι φυσικά σε παγκόσμιο επίπεδο να απαγορευτεί η αφαίρεση. Ε, προτείνουμε να εκφορτώνονται οι καρχαρίες ε, με τα πτερίγια άθικτα γιατί είναι ο απλούστερος και ο, ε, τρόπος, ο τρόπος και αυτός που εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε υψηλή γραφειοκρατία, υψηλό κόστος ως προς τα μέσα, το χρόνο, το ανθρώπινο προσωπικό που πρέπει να απασχολείται σε αυτό. Χρειαζόμαστε επίσης συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία κατά την εκφόρτωση, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επακριβώς τον πληθυσμό των καρχαριοειδών και να πάρουμε τις σχετικές αποφάσεις. Ε, ο κλάδος έχει εκφράσει ενσυχή σε σχέση με την αποθεματοποίηση. Ή πρότειναν βέβαια εν μέρη να τεμαχιστούν τα τερίγια και να διπλωθούν. Ε, σας ε, είπα ότι ορισμένες χώρες ε, το επιτρέπουν, άλλες παλαιόγια όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Παρίκα. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Γέρο. Gracias, señor presidente. Yo voy a seguir el consejo de la señora Patrao porque me parece que... Νομίζω ότι πράγματι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά γιατί όλοι έχουμε κάποιο συναισθηματισμό απέναντι στο θέμα, αλλά πρέπει να δούμε ποιες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε στην πραγματικότητα. Και σύμφωνα με όσα άκουσα, άκουσα διάφορους πρωταγωνιστές, ενδιαφερόμενα μέρη, συλλογικότητες που ανησυχούν για την πρόταση της Κομισιόν και κατόπιν άκουσα και εσά. Μου φαίνεται ότι τα είπατε με πάρα πολύ ακρίβεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρει αντίρρηση κανείς στα δικά σα ε, επιχειρήματα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι η Κομισιόν βιάζεται εδώ ε, και θα μπορούσε κάποιος να φτάσει στο συμπέρασμα ότι εδώ δεν ε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, περισσότερο υπάρχουν υποψίες ότι δεν πληρείται και δεν γίνεται σεβασμακτός ο κανονισμός κυρίως. Αυτό το άρθρο 4 εγώ θα ήθελα να τροποποιηθεί γιατί οι εξαιρέσεις ε, πρέπει να είναι όσο δυνατόν λιγότερες και θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα για να γίνεται σεβαστός ο κανονισμός. Όμως, σε μένα απευθύνθηκαν ε, οικολογικές οργανώσεις που τους άκουσα πάρα πολύ προσοχή αλλά μην προκνοείτε ότι γι' αυτό το λόγο θα έχω την τάδε τη δίνα θέση. Αυτοί στράφηκαν σε μένα και επίση απευθύνθηκαν και σε άλλε συναδέλφου. Και δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ άκουσα τι οικολογικέ οργανώσει πρέπει να έχω την τάδε θέση, ενώ αν ακούσουν κάποιοι του πλειοκτήτε θα έχουν άλλη θέση. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να αφήσουμε τι προκαταλήψει κατά μέρου και να σκεφτούμε τι διακυβεύεται. Αυτό που διακυβεύεται είναι ότι υπάρχει μια αμφιβολία που κάποιοι θεωρούν ε, ότι είναι λογική και κάποιοι όλοι για το αν υλοποιείται αυτή η πρακτική, όχι δηλαδή. Και πέρα από την ηθική σκοπιά, ε, έχουμε και κάποιες αξίες που περισπίζουμε στην Ευρώπη και επομένω πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για να ε, ρυθμίσουμε το θέμα αυτό έτσι ώστε τα σκάφη που ε, αλλιεύουν αυτό το είδος να το κάνουμε το σωστό τρόπο. Γιατί τελικά όταν ε, φτάνουμε στην εκφόρτωση βλέπουμε ότι αν είναι δυνατόν ε, να, να συνοδεύεται ε, από τα πτερίγια ο Καρχαρία το σώμα του Καρχαρία και η απόψυξη να γίνεται ταυτόχρονα έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί να γίνει διαφορετική θέση σε εμπορία των πτεριών και του σώματος. Και έτσι δεν θα έχουμε καμία Ε, αυτή είναι μια πρόταση, υπάρχει και μια εναλλακτική πρόταση που άκουσα επί ε, την οποία και εγώ θα συμπαθούσα και θα ήταν να γίνεται ταυτόχρονη εκφόρτωση σε όλα τα λιμάνια των πτεργείων και των σωμάτων. Έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι, γιατί ποτέ δεν θα είμαστε 100% σίγουροι, εκτός αν ψάξουμε στο βυθό της θάλασσας ε, να βρούμε το σώμα, το σφάγιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, εκτός αν είχαμε και έναν επιθεωρητή σε κάθε σκάφος. Βέβαια αυτό φαίνεται ότι οικονομικά δεν είναι και βιώσιμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε μία φόρμουλα που να μας δίνει την ασφάλεια, τη σιγουριά αυτού που υπερασπίζουμε επί της ουσίας. Γιατί αν ε, απλώς εδώ κινούμαστε βάσει της αξίας που δίνουμε στη ζωή κάποιων ζώων ακριβώς όπως θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τις σταυρομαχίες στην Ισπανία εγώ θα μπορούσα πολύ ξεκάθαρα να τοποθετηθώ αν μιλούσαν μόνο γι' αυτό. Όμως είναι πολύ πλοκό το θέμα. Αυτό το θέμα του ότι θίγει την Ισπανία και την Πορτογαλία, ναι μεν, αλλά υπάρχουν και αλεύματα που αφορούν άλλες χώρες περισσότερο. Αλλά τι να σας πω, ε, ουδής αναμάρτητος ή τέλος πάντων όποιος είναι αναμάρτητος πρώτος το λιθοβαλέτο. Και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την αρχή και να μην απομακρύνονται τα πτερίγια από τους καρχαρίες. Νομίζω ότι λοιπόν καλό θα ήταν να πάρουμε τον απαραίτητο χρόνο να εργαστούμε και ε, να μην ε, εγκρίνουμε ε, την πρόταση της Κομισιόν, τουλάχιστον το αιτιολογικό εγώ δεν θα ήθελα να το εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εγώ, όχι, ο κύριος Σάντσες μάλλον. εγώ θα ήθελα να σας πω ότι το φίνινγκ είναι μια απαγόρευση που είμαστε βρίσκει απόλυτα σύμφωνους ε, και νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε και τη βιωσιμότητα του Καρχαρία, αλλά πέραν αυτού θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θετούμε και λογικά μέτρα, μέτρα ελέγχου, θνηλασιμότητας, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε να ε, επιβάλλουμε και υπερβολικά έξοδα στο στόλο μας. Δηλαδή, ε, το να γίνεται μια διαδικασία επί του σκάφους ε, σημαίνει ότι υπάρχει και ένα κόστος και ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλες απαιτήσει όπως κανόνες προέλευσης κτλ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι λογικό να πρέπει να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής για να αποφύγουμε τα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλικία, αν κατάλαβα καλά, από ό,τι κατάλαβα θα μπορούσαμε να έχουμε επιπτώσει 40 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο μήνα στην ε, Γαλλική, ότι περνούν το χάρη υπήρχε το 2011 αύξηση 20% της αλίας ε, στην και 3.000 ε, ε, άτομα εθίγησαν από κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι είναι λογικό να εργαστούμε ως προς το να βελτιώσουμε τους ελέγχους και την χρησιμότητα και να έχουμε και μία περίοδο μεταβατική έτσι ώστε ο στόλος που ελεύει ψάρια να μπορεί να τα εκφορτώνει ε, μαζί και τα πλοία κατάψυξη να εκφορτώνουν ξεχωριστό και αν πρέπει να έχουμε ελέγχους να λάβουμε τα ανάλογα μέτρα. Γιατί είναι βιώσιμη η βιωσιμότητα των καργαριών με την ανάπτυξη του ελευτικού μας κλάδο. Νομίζω ότι αν το σκεφτούμε διαφορετικά θα ήταν παράλογο και μη υπεύθυνο. Μάλιστα, ευχαριστούμε στον τον κύριο Πρεσέδο. Ε, Πρόσφαση. Ε, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήδη συζητήσαμε διαμακρών σήμερα. Να πω καταρχήν ότι είμαι πεπισμένος ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα από την κυρία Πρατράουνεβε, την κυρία Φράγκα και ίσως κάποιους ακόμη ευρωβουλευτές. Και αυτά, αυτές οι λύσεις υπάρχουν και περιγράφονται διεξοδικά στη μελέτη αντικτύπου, στην αξιολόγηση αντικτύπου και αλλού γιατί αναζωπηρώθηκε η συζήτηση μετά την δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης αντιχτύπου και ήδη τρεις φορές στο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου το συζητήσαμε, μια φορά το συζητήσαμε και στην ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με εμπειρογνώμονες που είναι μάλιστα εδώ και αντιπροσωπεύουν τον τομέα. Για τρεις ώρες το συζητούσαμε. Δηλαδή πια μπήκαμε σχεδόν σε κάθε λεπτομέρεια. Μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις νομίζω ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις που θα λύσουν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζει ο κλάδος, θέματα εμπορίας, υγιεινής, ποιότητας, αποθήκευσης, ασφάλειας και ό,τι άλλο μπορεί να μην ανέφερα αυτή τη στιγμή. Να υπογραμμίσω ότι παρά την ανησυχία ότι μπορεί με όλα αυτά να θέσουμε σε μειονεκτική θέση τον ευρωπαϊκό κλάδο, εφιστώ την προσοχή στην νομοθεσία που υπάρχει ήδη σε άλλες χώρες στον κόσμο. Κάποιες χώρες από αυτές ήδη αναφέρθηκαν εδώ, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν 8 χώρες Κεντρικής Αμερικής που έχουν πολιτική για να μένουν εκεί τα πτερίγια. Υπάρχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ταϊβάν, και το υπογραμμίζω γιατί είναι μια χώρα μεγάλη ως κέντρο μεταποίησης και αλίευσης Καρχαρία και είναι μια χώρα που την αναφέρομαι ως ε, την πλέον υπέτειο χώρα για το φίνινγκ αυτό. Τώρα έχουν πολιτική που ε, προβλέπει την προσκόλληση παραμονή των πτερυγίων. Υπάρχουν λοιπόν τώρα ε, στοιχεία η συζήτηση αυτή έγινε και στους, στις ΠΟΔΑ. Τις επόμενες μέρες ε, θα γίνει η συνεδρίαση ε, της Επιτροπής για τον Τόνο και θα υπάρξουν ε, ε τροποποίησεις της νομοθεσίας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι φόβοι ότι θα υπάρξουν μειονεκτήματα από την πρώτη πρόταση της Κομισιόν δεν φαίνεται να ευσταθούν. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι αυτή η αναλογία του 5%. Η προβληματική της αναλογίας του 5% περιγράφεται διεξοδικά στην αξιολόγηση αντικτύπου. Θέλω όμως να ρωτήσω σε αυτό το σημείο τι κάνουν άλλοι τομείς, τι κάνουν τα σκάφη ψυγή άλλων χωρών όταν θα πρέπει να τηρήσουν ε, αυτή την αναλογία 5%. Ψαρεύουν διαφορετικά είδη καρχαριών, πουλάνε σε διαφορετικές αγορές, μεταποιούν διαφορετικά. Μου είπαν ότι κάποιοι στόλοι δεν διατηρούν όλα τα πτερήγια όπως οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Αλλά δυσκολεύομαι να το, πιστεύω, να το πιστέψω αυτό γιατί έχουν μεγάλη αξία τα πτερήγια και η τελική αγορά είναι η ίδια αγορά. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να πετούν λοιπόν πτερήγια καρχαριών όταν αυτά αξίζουν πολλά λεφτά και στην ασιατική αγορά που πάνε μιλάμε για ε, εκατοντάδες ευρώ ε, το κιλό. Μπορεί στην ασιατική αγορά. Μπορεί στην εκφόρτωση τη τιμή να είναι 12-15, αλλά εκατοντάδες ευρώ στοιχίζει στην αγορά. Αν, άλλοι, ε, ε, αν το δούμε πώς ε, τηρούν την αναλογία και τι κάνουν, θα είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω, ε, ε, δεν, επιμένει η Κομισιόν σε σχέση με την, ε, το ζήτημα της αναλογίας. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι μια πολιτική παραμονή των πτεργίων στο σώμα. Τώρα, για τα στατιστικά στοιχεία και το έγγραφο με τα στατιστικά, έχουμε δει ένα έγγραφο που μας το έδωσαν οι Ισπανικές αρχές και το συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου αλλά και διμερώς με το Ισπανικό Υπουργείο. Είναι σύνθετο το έγγραφο αυτό. Ένα, μία από τις ανησυχίες που ακούσαμε σήμερα είναι να αποφύγουμε, να φορτώσουμε περισσότερο τον τομέα και να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Το έγγραφο που προτείνεται ε, πραγματικά όμως ε, ε, είναι η επιτομή του περισσότερου φορτίου, γιατί θέλει πολύ μεγάλα και δύσκολα συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου με πολλές φραγίδες και πολλές από τις φραγίδες ε, θα πρέπει να δοθούν από λιμάνια τρίτων χωρών πριν φτάσει στο, το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Ισπανικές αρχές μας είπαν ότι δεν έχουν καν εμπιστοσύνη ε, στο, στην αξία της φραγίδας. Τι σημαίνει, ποιος ε, επιθεώρησε, ποιος φράγισε το έγγραφο. Πιστεύω λοιπόν ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι ιδεώδης λύση. Εις ό,τι αφορά τις άδειε και τον αριθμό των αδειών που εκδίδονται, αυτό κυμαίνεται ετησίως. Είναι περίπου 200. Δεν μπορώ να σας πω πόσες ήταν πέρσι, γιατί δεν πήραμε ακόμα τις εκθέσεις για την περσινή χρονιά αλλά ο πορτογαλικός αριθμός ήταν μεταξύ 11 και 49 τα χρόνια 2004 με 2010 και ο ισπανικός αριθμός αδειών κοιμάνθηκε μεταξύ 164 και 200. Τώρα μας λένε 141, ίσως είναι ένα πρόσφατο στοιχείο που ακόμα δεν έφτασε στα χέρια μας. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, να κάνω ένα σχόλιο. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γκαρσία, κυρίως, ε, που είπε ότι βιάζεται πολύ η Κομισιόν. Όχι. Τίποτε το βεβαιασμένο δεν υπάρχει στην πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν στηρίχθηκε σε πολύ διεξοδική μελέτη αντικτύπου. Ε, επί χρόνια συζητείται ε, ε, προηγήθηκαν ευρύτατες διαβουλεύσεις και αντιπροσωπεύονται διεθνείς τάσεις στην επιστήμη, ε, οι απόψεις των πόδα κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πατράου, για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι, αλλά θα πω ότι σε σχέση με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Έχουμε ήδη συζητήσει με εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν επικοδομητικό ο διάλογο, αλλά αυτά που άκουσα σήμερα τώρα με αφήνουν άναυδη. Ε, εντοπίζουν την συζήτηση γύρω από τις υποψίες παραβίασης. Ε, δηλαδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι γίνονται κάποια πράγματα στην Πορτογαλία και κανείς δεν είδε ποτέ ούτε άκουσε τίποτα. Μα δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις υπόνες υποψίες για να κάνουμε διάλογο. Δεν ξέρω τι να σας πω μετά. Ε, ποιος θα προτάξει το αντεπιχείρημα, έτσι, ποιος θα δώσει τον αντίλογο. Επίσης, ε, τι είναι αυτές οι προκαταλήψεις για τον ε, τομέα, γιατί μας λέτε ότι δεν είναι μεγάλος. Ε, λοιπόν, ε, ας σταματήσουμε. Ε, μετά μας μιλήσατε για την έκθεση αντικτύπου λοιπά. Μα συγγνώμη, εγώ σας δίνω στατιστικά στοιχεία και σας λέω ότι θέλουμε να απαλείψουμε τις υποψίες σε σχέση με την αφαίρεση των πτερυγίων. Μετά μου λέτε ότι είναι περίπλοκα τα στατιστικά στοιχεία και λυπούμαστε εμεί στον κλάδο επειδή δεν μπορεί να διαβάσει τα περίπλοκα στατιστικά στοιχεία. Μα ε, σοβαροί είμαστε, δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Ε, λέτε ότι υπάρχουν πρακτικές ε, λύσεις. Για όλα μας λέτε κύριε Ντέιβες. Ε, λοιπόν, δε, γιατί είμαστε εδώ πέρα αν υπήρχαν οι λύσεις, δηλαδή τι είναι, ανόητοι όλοι στον αλληλευτικό κλάδο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν μπορούν να βρουν τις λύσεις, ε, δεν, καταλαβαίνω περί τι πρόκειται. Αξιότιμοι συνάδελφοι, έκανα μία εισαγωγική παρουσίαση, σας ε, εξέθεσα τα ερίσματα της σκέψης μου και σας είπα ότι θα έχω ανοιχτό πνεύμα, δεν θέλω να είμαστε προκατά προκαταλημένη και να ε, ε, ισχυριζόμαστε ότι καμία μη κυβερνητική ε, δεν έχει στοιχεία. Εγώ με όσε πρόσωπο του κλάδου μίλησα, με παρέπιζαν σε 5-6 διαφορετικές ΜΚΟ που υποστηρίζουν αυτή την θέση. Οπότε Γι' αυτό σας λέω ότι ας αφήσουμε τις ε, προκαταλήψεις, ας αφήσουμε τις απλοϊκές ε, λύσεις. Χρειαζόμαστε τις πλέον πρόσφορες ε, λύσεις. Εμείς θέλουμε τις πλέον κατάλληλες λύσεις, όχι τις απλούστερες λύσεις. Θέλουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα που διακυβεύονται. Θέλουμε να επιλύσουμε τις διαφορές που υπάρχουν για αυτό το θέμα σε αυτό το πλαίσιο έκανα εγώ συγκεκριμένες ε, προτάσεις και πρέπει να σας πω ότι ε, οι πρώτοι συνάδελφοι που πήραν το λόγο ούτε καν αναφέρθηκαν στις δικές μου προτάσεις, αυτό που θα θεωρούσα εγώ ως εισηγήτρια, καλή συμβαστική λύση, ότως ώστε να ε, βρούμε μαζί ε, την ε, ε, κατάλληλη λύση και όχι να ξεκινάμε όλοι με τις προκαταλήψεις μας. Τέλο εγώ σας έχω παρουσιάσει κάποιες προτάσεις, αλλά δεν είναι και βίβλος, έτσι, θα τις τροποποιήσω. Εάν μου δώσετε άλλα στοιχεία, αν τροφοδοτήσετε με σκέψεις σας τη συζήτηση, θα, μαζί σας θα βρω τη συνετική λύση. Δεν προτείνω έτοιμες λύσεις ένα αυτό. Τώρα, το να μου λέτε ότι υπερασπίζομαι το εθνικό συμφέρον, μα τι λέτε, ε, γιατί είμαστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα ε, ε, θέλουμε να υπερασπιστούμε την, ε, τον κλάδο ε, σε επίπεδο ένωσης, αλλά όχι εις βάρος του εθνικού κλάδου. σήμερα είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Λοιπόν, σε σχέση με τις αντίθετες πλευρές σε αυτή την συζήτηση. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά και... Θα πρέπει να βασιστούμε για να βγάλουμε μία άκρη στις αρχές που πρέπει να διέπουν τη δράση μας. Ποιες είναι αυτές. Η δική μου αρχή, όπως σας είπα και στην πρώτη παρουσίαση, είναι πρώτον να αναγνωρίσουμε όπως όλοι αναγνωρίζουν. Α, ναι, και παρεπιπτόντως, ε, ε, ε, όπως είπε η κυρία Φράγα, δεν υπάρχουν, λέει, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δίνουν στοιχεία και ότι υπάρχουν μόνο υπόνοιες. Αυτό μας είπε. Μάλιστα, ναι, τι να κάνουμε, όμως υπάρχουν υποψίες. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να επισκιάζεται ο στόλος μας από αυτές τις υποψίες και γι' αυτό ε, εισηγούμε λύσεις, όχι ριζοσπαστικές. Ε, και όχι ριζοσπαστικέ, γιατί πρώτον είναι μόνο πόνοιε, ε, και δεύτερον και επιμένω ε, εφόσον κάνουμε τη μεταρρύθμιση και εφόσον μπορεί να πληγούν στόλοι δύο χωρών και μελλοντικά ίσως και περισσότερων, μα τι να κάνουμε, είναι κράτη-μέλη της Ένωσης, έτσι, η Ισπανία και η Πορτογαλία και τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν τα συμφέροντα του στόλου του ευρωπαϊκού από τη μία και του ισπανοπορτογαλικού και να βρούνε μία ισορροπία. Είναι ουσιαστικές οι ζημιές τις οποίες αναφερόμουν και όπως είπε και η συνάδελφος έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία από τη Γαλλική. Ε. Θα σας δώσουμε και άλλα. Είμαστε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ακόμη. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι τίθεται ζήτημα ζημιών ε, και αυτή η μεταρρύθμιση θα επισύρει και άλλες επιπρόσθετες ζημιές, ε, οπότε δεν μπορείτε να μου λέτε ε, ότι προδικάζουμε. Συγγνώμη, ε, υπάρχουν υπόνοιες, υπάρχει βάση. Χρειαζόμαστε χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για να συλλέξουμε στοιχεία και για να προσαρμοστεί ο στόλος στη μεταρρύθμιση και όχι να πυρπολείται διαρκώς με προτάσεις που είναι επιζήμιες για τον κλάδο. θα ήθελα ε, να ε, αναφερθώ σε κάποια αντιφατικά σημεία, παρεμβάσει των συναδέλφων. Είπανε δεν υπάρχει τεκμηρίωση των ζημιών και ως εκ τούτου δεν αξίζει να το συζητάμε. Εγώ λοιπόν ε, ε, προσθέτω ότι δεν θα μιλάγαμε καν για το φίνινγκ άμα δεν υπήρχαν ε, ε, υποψίες. Εντάξει, υποψίες όμως υπάρχουν, στοιχεία δεν έχουμε, το ξαναλέω αν λέμε το πτερίγιο θα παραμείνει ε, στον κορμό ή θα αφαιρεθεί κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα επιμέρους σημεία. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει θέληση διαλόγου και με τα στοιχεία που έχουμε να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε λύση. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους στοιχεία που δεν συζητήθηκαν καν εδώ αν ή μη τεμαχιστεί και αναδιπλωθεί το περίγειο δίπλα στο σώμα, βάσει της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να φτάσει στις αγορές υπό αυτή την μορφή, τι σημαίνει. Το ψάρι δεν μπορεί να Ε, μεταποιηθεί πρέπει να είναι ολόκληρο. Ε, όταν όμως γίνει η μερική απόψυξη στη συνέχεια για να αφαιρεθεί συνολικά το πτερίγιο πρέπει να αποψυχθεί τελείως ε, για να βγουν τα εντόστια του ψαριού. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς ο εξπλαχνισμός πρέπει να γίνεται ε, πάνω στο πλοίο. Γι' αυτό σα λέω, πρέπει όλοι να έχουμε ανοιχτό πνεύμα, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν συζήτησαν και μην ξεχνάτε και έναν άλλο σημαντικό παράγοντα. Όταν κάνουμε του υπολογισμού, και θα σα τα πω αύριο, γιατί το έγγραφο εργασία αύριο θα μεταφραστεί, δεν εξαντλεί βέβαια όλη την επιχειρηματολογία. Έγγραφο εργασία είναι, το λέει και το όνομά του. Θα μετεξελιχθεί, αλλά θα δείτε ότι ε, όταν μιλάμε για γλαυκοκαρχαρία 200 κιλών, η αξία πώληση του κορμού υπερβαίνει την εμπορική αξία των πτερυγίων. Άρα για ποιο λόγο να γίνεται το φινί, για ποιο λόγο να έχουμε μόνο τον κορμό, δεν, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Ή αλλιώς, τι να πω, θεωρώ, θεωρούμε ότι είναι ηλίθιοι όλοι στο, στον αλληλευτικό κλάδο και δεν ξέρουν, ε, δεν γνωρίζουν άλλη λύση. οι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν με εμένα για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, να συζητήσουν για τα στοιχεία κτλ. Ε, είναι ευπρόσδεκτοι. Και εγώ ίδια θα έρθω σε επαφή με όλου του κοιόντες, ε, διότι έγιναν συγκεκριμένε ε, προτάσει, αλλά δυστυχώ ούτε καν τι χρησιμοποίησαν οι συνάδελφοι για το διάλογο. τέλο πάντων, υπάρχουν στοιχεία σημαντικά όπως αυτό της ίχνη λασιμότητας, ε, δηλαδή αν εκφορτωθούν σε διαφορετικά λιμάνια και διαφορετικές χρονικές στιγμές ο κορμός και τα πτερίγια, ποια ίχνη λασιμότητα, για ποια ίχνη λασιμότητα μιλάμε. Νομίζω κακή τύποι στη Μιλάνε ε, κάποιοι όταν μας λένε ότι πρέπει να επιτρέπεται αυτό. Ε, και τα ίδια ε, για τους στόλους ε, νοπών σε, κατά τη διαστολή με τους στόλους των κατεψυγμένων. Αυτά τα επιχειρήματα δεν ευσταθούν κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστούμε κύριε Πατρά. Μάλιστα θα περάσουμε τώρα στο σημείο 5 τροπήση του κανονισμού για θέσπιση σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Κανονισμό 302 του 2009 στι 20 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε στην ε, Επιτροπή Έκθεση και ε, προσπάθησε ο εισηγητής ε, να καταλήξει σε μια πρώτη ε, συμφωνία ε, και στις 9 Φεβρουαρίου έγινε ο τριμερής διάλογος και εκεί Γίνανε δεκτά όλα τα σημεία που παρουσίασε το Κοινοβούλιο, εκτό από τρει ε, συγκεκριμένα, τρεις συγκεκριμένα θέματα που προτάθηκαν από το Συμβούλιο, όπου ζητάει η Κομισιόν να εθετηθούν εφαρμοστικές πράξεις ε, σε ό,τι αφορά το άρθρο 1.9, δηλαδή τη μεταβίβαση της ε, πράξης ε, σε κλουβιά, το άρθρο 1.10 και τα μητρώα πληροφοριών. Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ λεπτομερείς οι κανόνες και ότι δεν χρειάζονται περιπτέρω ανάπτυξη και καθώς δεν κατέληξε κάπου τριμμένης διάλογος, σταμάτησε έτσι ώστε να μπορέσει να ε, καταλήξει σε μία θέση το Κοινοβούλιο, γιατί δεν είχε καθορισμένη θέση. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε τώρα, για να υπάρχει μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ορισμένε πτυχέ όπου δεν είχε ληφθεί απόφαση. Και χωρί περαιτέρω θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα και σε όσου υπόλοιπου θέλουν να τοποθετηθούν στη συνέχεια. Κύριε Ρωμέβα, πολύ καλά τα εξήγησε ο Πρόεδρος, το θέμα είναι ακριβώς έτσι. Όταν εμείς ε, συνεδριάσαμε στον τριμερή διάλογο, είχαμε μια σαφή εντολή, ναι, στην περίπτωση μου συζητή και οι σκιώδει είχαμε σαφή εντολή από του συναδέλφους για ορισμένα σημεία. Τα σημεία αυτά είναι αυτά από τα οποία είχαμε εντολή και μπορέσαμε να τα διαχειριστούμε και υπήρξε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Και έτσι λοιπόν ε, προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. μπορεί να περάσει στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια, όμως παρουσιάστηκαν τρία θέματα πράγματι, τα οποία είναι σημαντικά. Πρόκειται για ένα θέμα σε τρία μέρη, για να το πω έτσι, γιατί το ουσιαστικό θέμα είναι το ίδιο, αλλά υπάρχουν ε, τρία διαφορετικά παραδείγματα. Έχουμε το θέμα της ε, χρήσης ήμις ε, των εκτελεστικών πράξεων για να ζητήσουμε από την Κομισιόν για να αποφασίσει σε ορισμένες περιπτώσεις ε, να μας πει πώς θα εφαρμόσουμε τον κανονισμό σε ορισμένα από αυτά τα τρία σημεία. Οι τρεις πτυχές που αναφέρθηκαν ήταν καταρχήν ε, το θέμα όσα έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της ε, μεταφόρτωσης, τη μεταφοράς δηλαδή από το δίκτυ πώς μεταφέρεται στο κλουβί. Και το δεύτερο θέμα αφορούσε τεχνικά ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν να κάνουν με ε, το τι απαιτείται στον κανονισμό ICAT και και όχι τόσο το Συμβούλιο, μάλλον ε, όχι μόνο ακριβώς το Συμβούλιο, αλλά κάποιο κράτος μέλος θέση το θέμα για το πώς γίνεται ο υπολογισμός ε, και η διευκρίνηση των στοιχείων την ε, στιγμή που μπαίνουν στο κλειδιά ορισμένα αλλιεύματα. Μεθοδολογία λοιπόν υπολογισμού και εκτίμηση ορισμένων αλλιευμάτων και υπήρξε και ένα θέμα το οποίο είναι πιο σχετικό με τις παγίδες. Και πάλι υπήρχε θέμα με τις πληροφορίες και τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών και φαινόταν ότι κάποιο κράτος μέλος δεν είχε καταλάβει πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Στη συζήτηση που είχαμε το Συμβούλιο διατήρησε τη θέση του. Δηλαδή, ε, ήθελε να υπάρχουν εφαρμοστικέ πράξεις, ενώ η Κομισιόν διατηρούσε τη θέση της, που θεωρούσε ότι δεν είναι απαραίτητο και μάλιστα το αντίθετο, ότι θα μπορούσε να υπάρξει καθυστέρηση στη διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού και θα μπορούσε αυτό να έχει και συνέπεια για ε, την παρουσίαση, τη λογοδοσία που πρέπει να κάνει στη συνέχεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ICAT. Δεν είχαμε κοινή θέση και αποφασίσαμε λοιπόν να επανέλθουμε εδώ στην Επιτροπή για να μπορέσουμε να δούμε με τους συναδέλφους ποια θέση πρέπει να πάρουμε ως Επιτροπή Αλίας. Καθώς ε, μεταξύ μας ε, στην Κομισιόν, καθώς είμαστε εδώ και έχουμε ε, εκπροσώπους και από Κομισιόν και το Συμβούλιο, θα πρέπει να τους ακούσουμε όλους. Εγώ έχω τη δική μου θέση. Νομίζω ότι η Επιτροπή έχει δίκιο. Και έχουμε τα δύο θέματα. Τα τεχνικά ζητήματα που τέθηκαν από ορισμένα κράτη-μέλη μπορούν να επιληθούν. Βασικά, διμερός. Δεν υπάρχει δηλαδή περαιτέρω πρόβλημα. Και δεύτερον, ο κίνδυνος ε, που θα υπέθετε το να έχουμε προηγούμενο, ε, επιμένω, έχει να κάνει με τον ερθρό τόνο και θα μπορούσαμε να καταστήσουμε πιο δύσκολο το ρόλο της Κομισιόν τη στιγμή της διαχείρισης της εντολής που της δίνεται από τα κράτη-μέλη στο ICAT. Δηλαδή, ε, αν ε, η Κομισιόν ε, βρει ότι δεν υπάρχει σαφής λύση ή ότι είμαστε ακόμα σε ε, διαδικασία συζήτηση ε, θα μπορούσαμε να έχουμε το εξή αποτέλεσμα και το είδαμε αυτό. Στι φορέ θα μπορούσε από την πλευρά του ΆΙΚΑ να σταλεί μια προειδοποιητική επιστολή και αυτό θα έχει επίπτωση όχι μόνο στι ποσοστώσεις αυτού του συγκεκριμένου κράτου μελού, αλλά στι ποσοστώσεις όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ κατανοώ ότι είναι πρόβλημα κοινό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι εγώ θεωρώ ότι η πρόταση τη Κομισιόν είναι λογική και κάτι παραπάνω από λογική και εγώ ω αυτή προτείνω όμως ε, ίσως να υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορεί να διαφωνούν. Γι' αυτό το θέτω εδώ προς συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριο ε, Στίβενσον, κυρία Φράγκο και κατόπιν εκπρόσωπη Συμβουλή του Κομισιόν. Παρακαλώ, Στίβενσον. Thanks, <coughs> President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Just cut to the chase and, Ας μπούμε στο θέμα και ας διευκρινίσουμε τι ε, περί πρόκειται. Αν ακολουθήσουμε την σύσταση του Συμβουλίου για τον Ερυθρό Τόνο, σε αυτά τα τρία σημεία θα καθυστερήσουμε την ε, εφαρμογή του κανονισμού και θα περάσει και άλλη μια περίοδος ε, που δεν θα ρυθμίζεται η αλία του τόνου. Αυτό το παιχνίδι παίζει το Συμβούλιο εμείς δεν είμαστε ανόητοι, ξέρουμε ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι και όταν ακούω ότι ένα, ε, μια εφαρμοστική πράξη προβλέπει ότι θα τους ενημερώνουν για το πότε θα ε, ε αρχίζει να λειτουργεί φωτογραφική μηχανή για να παρακολουθεί τα, τους νεαρούς τόνους που μπαίνουν στους κλοβούς. Ε, τι, να πω, ε, δεν μας σέβονται. Εγώ υπέθετα ότι η Κομισιόν θα ζητάει στα πλαίσια της συνθήκης και όχι το Συμβούλιο εφαρμοστικές πράξεις. Θα πρέπει να πει στο Συμβούλιο ότι θέλουμε εφαρμοστικές πράξεις. Γι' αυτό άρχισα να έχω υποψίες ότι παίζονται παιχνίδια εδώ που εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να τα παίξω χρειάζεται το απόθεμα του ερυθρού να προστατευτεί και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να περάσει κι άλλη περίοδος ασίδωτης αλληλείας που θα καταστρέφει το απόθεμα. Κυρία Φράγκα. Ευχαριστούμε κυρία Φράγκα. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί όλα τα σημαντικά θέματα έχουν επιληθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αλλά να πω ένα παράπονο. Αισθάνομαι ότι στην ε, συνάντηση του τριμερού διαλόγου ήμουν μόνο εγώ και ο συγητής και καθώ εγώ είχα άλλη θέση και ο συγητή, άλλοι δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου. Και θα ήθελα να μην ξαναγίνει αυτό στο μέλλον, ε, γιατί αν ε, οι σκιώδει συγητέ δεν έρχονται στου τριμερού διαλόγου, σε αυτέ τι καταστάσει καταλήγουμε που είναι παράλογε. Τώρα, πέρα από αυτό, εγώ είχα την αντίθετη θέση ε, αυτή που εξήγησε ο κ. λόγω του εξή. Αυτή η θέση να ζητήσουμε να εφαρμόζεται το άρθρο 291 για τα άρθρα 22, 24, 26 είναι άρθρα πάρα πολύ τεχνικά αυτά και μιλάμε για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο είδος όπως είναι ο ερυθρός τόνος και ε, όλα τα κράτη-μέλη που αλλιεύουν ερυθρό τόνο έχουν προβλέψει τη δυνατότητα και έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ε, αυτή η ερμηνεία, η τόσο τεχνική, να μπορεί να είναι ε, απαραίτητο να εφαρμοστεί μέσω εκτελεστικής πράξης έτσι ώστε να έχουμε την ίδια ερμηνεία για όλους. Και τα κράτη-μέλη δεν είπαν να είναι υποχρεωτικό όλα αυτά να μεταφραστούν σε εκτελεστική πράξη. Λένε may Δηλαδή, η Κομισιόν, αν κάποια φορά θεωρήσει απαραίτητο σε συμφωνία με τα κρατημέλη ότι θα πρέπει να υπάρχει εκτελεστική πράξη, τότε η Κομισιόν που έχει την πρωτοβουλία θα μπορέσει να θέσει μια εκτελεστική πράξη. Και εγώ νομίζω ότι θα μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη δυνατότητα ανοιχτή, ε, καθώς και την πρωτοβουλία την έχει η Κομισιόν, δεν βλέπω να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει επίπτωση στι ποσοστώσει κτλ. Αυτή είναι απλώ η δυνατότητα κάποια συγκεκριμένη στιγμή, γιατί έχουμε ΜΕΙ και όχι ΣΑΛ και το επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι η πρωτοβουλία τη Κομισιόν. Η Κομισιόν ε, κάποια στιγμή, αν το κρίνει απαραίτητο, αφήνει αυτή την πόρτα ανοιχτή δηλαδή. Απλώς αφήνουμε μία πόρτα ανοιχτή ε, εφόσον χρειαστεί. Κύριε Στίβενσον, αν εγκριθεί αυτό δεν ε, αντίκειται στην εφαρμογή κάποιου μέτρου, Απλώ αφήνουμε ανοιχτή τη δυνατότητα στην Κομισιόν κάποια συγκεκριμένη στιγμή να προβεί σε εκτελεστική πράξη για αυτά τα τρία άρθρα, αν χρειαστεί σα ξαναλέω. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω ούτε καν ε, την Κομισιόν γιατί θέλει να κλείσει την πόρτα. Γιατί να θέλει να κλείσει την πόρτα αν ε, μπορεί να το κάνει αυτό κάποια στιγμή. Αν δεν θέλει δεν κάνει, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. βίντεο. φαίνεται παράλογο όμως να κλείσει την πόρτα η Κομισιόν, ε, γιατί η νομική υπηρεσία είπε ότι μιλάμε για εκπληστική πράξη, τίποτα άλλο δεν είναι. Αυτό ζήτησαν τα κρατη Έτσι λοιπόν, αν συμφωνείτε με την πρόταση, μπορείτε να βάλετε The Commission may adopt implementing acts as regards κτλ. Δηλαδή, να αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Δεν dejarla abierta, por si en un momento dado esto es κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλη την εργασία που έχει γίνει για αυτό το θέμα που είναι πολύ σύνθετο. Για τις εργασίες, λοιπόν, και του Κοινοβουλίου ε, και των, ε, της Τωρινής και της προηγούμενης Προεδρίας. Ε, είναι όπως ε, ανέφεραν και ε, οι προλαλήσαντες, τεχνικό, δύσκολο το ζήτημα και ε, ιδιαίτερα ευαίσθητο λεπτό διότι ε, είναι εμβληματικό το είδος και ο φάκελος ο ίδιος για κάποια κράτη-μέλη. Ε, Παρ' όλα αυτά καταλήξαμε σε μια συμφωνία για σχεδόν όλα τα επιμέρους σημεία του εγγράφου ε, εργασίας. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα που υπάρχει ακόμη διαφωνία. Δεν είναι όμω τεχνικά ζητήματα. Σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματο και προκειμένου, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, σχετίζονται με την αλληλευτική περίοδο του 2012. Ήδη έληξε η προηγούμενη του 2011 χωρί να έχουμε ένα νομικό εργαλείο μεταγραφής στην εθνική νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν ένα νομικό πρόβλημα και προσπαθούμε κατά περίπτωση να το λύσουμε σε συνεργασία με τα συμβαλόμενα μέρη επιθυμούμε σε κάθε περίπτωση πρωτού αρχίσει η αλευτική περίοδος 2012 ε, να έχει ρυθμιστεί το ζήτημα. Είναι δε πάρα πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί διότι οι οικονομικοί φορείς που ενδεχομένω θα πληγούν από αυτό το θέμα έχουν ήδη σχεδόν αρχίσει την δραστηριότητά τους. Είμαστε σε προκεχωρημένο στάδιο προετοιμασίας της αλληλευτικής περίοδου του 2012 ε, και ε, ε, ο Μάιος Ιούνιος το, η περίοδος εχμής αν θέλετε για την αλλιευτική περίοδο και είμαστε ήδη τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου προετοιμάζονται όλοι για αυτή την περίοδο εχμής και τα ελεγκτικά όργανα, ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών πρέπει επίσης να προετοιμαστούν για να εκπονήσουμε τα ελεγκτικά μέτρα. Είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο, το ξαναλέω και επιμένω ότι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το να μην διαθέτουμε ένα τέτοιο νομικό εργαλείο για τόσο σημαντική ελευτική περίοδο όπως το 2012 θα ήταν κάτι που σαφέστατα θα δημιουργούσε πρόβλημα όπερ και θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία ε, ως προς ε, την συνεδρίαση αυτής της χρονιάς και φυσικά ως προς την αλληλευτική περίοδο. Αυτά για το χρονοδιάγραμμα ε, της ε, υλοποίησης και το γενικότερο χρονοδιάγραμμα. Δεύτερο σημείο. Η σύσταση ICAT είναι σαφής. Ε, ε όλες οι τεχνικές συζητήσεις έχουν ήδη ε, λάβει χώρα πρωτού αρχίσει μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες. Θεωρούμε επίσης ότι ε, υπό το φως των αποτελεσμάτων του πρώτου έτους ε, σε ισχύ αυτών των διατάξεων, έχουμε διαμορφώσει πλέον μια σχετικά ε, ξεκάθαρη εικόνα για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Λοιπόν, κατά την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, το να προετοιμάσει ένα νομοθέτημα σημαίνει απώλεια χρόνου και κάποιοι θα υποφεληθούν και θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο ως προς την εφαρμογή, ε, τη συμμόρφωση μάλλον ε, με τις υποχρεώσεις τους και υπενθυμίζω ότι το σύνολο των συμβαλωμένων μέρων στην ΑΕΚΑ θα εξετάσει αυτό το θέμα τον Νοέμβριο. Μας πιέζει ο χρόνος, ε, προκύπτει σαφώς από αυτά που σας λέω, οπότε όσοι έχουν τις υποχρεώσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς όμως τώρα τι γίνεται σε, εδώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατηρούμε την πάγια προσφορά μας. Δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές ε, και να συνεργάζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ούτω ώστε σε τεχνικό επίπεδο να εκπονήσουμε όχι εκτελεστικές ε, πράξεις, αλλά να προσφέρουμε μία ένα μεθοδολογικό προσανατολισμό, μια ε, μεθοδολογική κατευθυντήρια γραμμή. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα νομοθετήματα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά στη συνεργασία με εκπροσώπου άλλων θεσμικών οργάνων, με τον κλάδο, με του επαγγελματίε, με του επιστήμονε, ώστε να αναλύσουμε περαιτέρω να συγκεκριμενοποιήσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού. Καλούμε δε όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν να ε, συνεργαστούν μαζί μας, αλλά σας λέω ότι με αυτές τις εκτελεστικές πράξεις ε, το αποτέλεσμα ενώ θα καθυστερήσει η θέση σε ισχύ, ενώ πρέπει να συμβεί τώρα. Ε, Μάλιστα. Εκ μέρους του Συμβουλίου, κ. Chairman, Members of the committee. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, ως εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή που μου δίνει την ευκαιρία να σας απευθύνω άμεσα το ε, λόγο για να ε, παρουσιάσω τις απόψεις του Συμβουλίου. Όπως είπε ο, πρόεδρος, ο εισηγητής, ο κύριος ε, Ρωμέβα, με τον τριμερή διάλογο επετέφθη ο, πλήρη συμφωνία σχεδόν ε, για κάποιες τεχνικές τροπολογίες που θα διευκρινίσουν το σχέδιο της νομοθεσίας ε, που θα εφαρμόσει την σύσταση 10 κάθετος 04 της ΆΙΚΑΤ για το πολιετές σχέδιο ανασύστασης ε, στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Όπως όμως εξήγησε επίσης ο κύριος Ρωμέβα, Κάποια θέματα έπρεπε να παραπεμφθούν στην Επιτροπή σας για περαιτέρω εξέταση σήμερα. Τα άρθρα είναι τα άρθρα 22, 24 και 26 για να εξετάσετε εσείς. Εκεί το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να αναθέσει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Κομισιόν με βάση το άρθρο 291 της Συνθήκης. Το Συμβούλιο θεωρεί γενικότερα ότι σε σχέση με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν ότι οι νομοθέτες πρέπει να εξετάσουν την συγκεκριμένη κατάσταση εν προκειμένου και κατά περίπτωση και να αποφασίσει επ' αυτής της βάσεως αν οι νομοθέτες θέλουν ή όχι να αναθέσουν κάποιες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή επιτροπή ή καμιά φορά να μην τις αναθέσουν καμία αρμοδιότητα. Σε σχέση με τα ε, επίμαχα άρθρα, το Συμβούλιο θεωρεί ότι κάποια θέματα θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, ώστε να διασφαλίσουμε ε, αρμονική, ε, ομαλή εφαρμογή των κανόνων από όλους στην Ένωση. Η ΆΙΚΑΤ έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες, αλλά λίγα σε ορισμένα θέματα δεν είναι οι κανόνες απόλυτα σαφείς, γι' αυτό θέλαμε εκτελεστικές πράξεις. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες στον κλάδο, για να ξέρει ο κλάδος τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Επίσης σημαντικό είναι οι εθνικές ε, διοικήσεις να ελέγχουν, να επιθεωρούν σωστά, να επιβάλλουν τους κανόνες αν κάποιοι θέλουν να τους παραβιάσουν. Να εξηγήσω λεπτομερέστερα με παραδείγματα αυτό που εννοώ για το άρθρο 22 σχετικά με τις μεταφορές ε, λέει ότι ε, θα πρέπει να παρακολουθείτε η ε, απελευθέρωση στη θάλασσα με κάμερα του τόνου και θα πρέπει να δίνονται τα βίντεο στην γραμματεία της ICAT. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώνει η καταγραφή σε βίντεο και τι γίνεται με την ποιότητα. Επίσης για τον εγκλωβισμό υπάρχει ένα ε, ε, εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχει την ε, στιγμή του εγκλωβισμού. Θα πρέπει επίσης να δούμε το, την αναλογία του δείγματος που θα προβλέπετε και ποια θα είναι η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείτε. Για το άρθρο 26 σχετικά με την καταγραφή ε, του εγκλωβισμού και τις παγίδες. Υπάρχουν πολλές παγίδες, πάλι πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, αυτά είναι κάποια πρακτικά παραδείγματα που ελπίζω να βοηθούν να καταλάβετε την επιχειρηματολογία του Συμβουλίου. Και ε, τη θέση του σε σχέση με τι εκτελεστικέ πράξει ε, από την Κομισιόν. Σημειώνει το Συμβούλιο το γεγονό ότι η Κομισιόν δεν βλέπει ανάγκη για τέτοιε πράξει Γι' αυτό το Συμβούλιο προτείνει η Κομισιόν να μπορεί ενδεχομένω να εγκρίνει τέτοιε πράξει. Το Συμβούλιο αναμένει ότι καθ' αυτό εφαρμογή των κανόνων και τα πρακτικά προβλήματα που αναπόφευκτα θα ε, υπάρξουν θα δικαιώσουν το Συμβούλιο το οποίο πρότεινε τις ε, εκτελεστικές πράξεις και τονίζω ότι προφανώς η Κομισιόν λίγο μετά που τη θέσπιση το Νοέμβριο του 2010, τη θέσπιση της σύστασης από την ΆΙΚΑ, την ενημέρωσε ο, την ΆΙΚΑ το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τη σύσταση. Άρα λοιπόν τώρα ισχύει και εφαρμόζεται η σύσταση της ΆΙΚΑ. Και εδώ δεν πρόκειται για την ε, ε, μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Ε, το καλοκαίρι του 2011 ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι και οι κανόνες. Ε, ελπίζομαι και το Κοινοβούλιο θα συμμεριστεί τις απόψεις του Συμβουλίου, ούτω ώστε να υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση στην Κομισιόν. Κυρία Σάντσι Πρεσέδο, θα σας δώσω το λόγο, αλλά δεν μου το είχατε ζητήσει πριν. Δεν το ζήτησα ακριβώ ε, γιατί ήθελα να ακούσω τι είπαν η Κομισιόν και το Συμβούλιο, γι' αυτό δεν το ζήτησα. Λοιπόν, ε, σύμφωνα με τη συνθήκη, τα κράτα-μέλη είναι αυτά που είναι απευθεία υπεύθυνα για την εκτέλεση της ε, κοινωτικής νομοθεσίας και αυτό άλλαξε με τη συνθήκη της Λισαβόνα. Έτσι λοιπόν, ε, όταν τίθεται η αναγκαιότητα να υπάρχουν ε, κάποιες ομοιόμορφες προϋποθέσεις εφαρμογής ε, ή όταν υπάρχει αναγκαιότητα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να δίνει την ίδια ασφάλεια σε όλους και να μπορούμε να δείξουμε ότι στην Ευρώπη εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία και να διευκολύνουμε την Κομισιόν, μπορεί να είναι απαραίτητο να το θέσουμε ρητός, γιατί αν δεν τεθεί ρητός ότι η Κομισιόν μπορεί να προβεί σε εκτελεστικές πράξεις, δεν μπορεί να το κάνει η Κομισιόν και δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι είναι σημαντικό σε αυτό το θέμα να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη και θα πρέπει να το εγκρίνουμε και εμείς από την πλευρά μας. Και αυτή είναι μια απόφαση του νομοθέτη ούτως ή άλλως. Είναι ο νομοθέτης ο οποίος ε, καθορίζει πώς ε, πρέπει να εκτελεστούν ε, οι εντολές του. Έτσι λοιπόν οι νομοθέτες έχουν ένα λόγο και ζητούν από την Κομισιόν να έχει αυτές τις αρμοδιότητες και εγώ νομίζω ότι είναι λογικό κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να δεκτούμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κυρία Ρόντουστ. Oh, jetzt bin ich in Verlegenheit, weil ich meinem Νιώθω λίγο, αμήχαν... Νιώθω λίγο αμήχανη, γιατί δεν θέλω να φέρω αντίρρηση στο συνάδελφο. Ε, πάντως, εμείς θέλαμε κάτι εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικές πράξεις. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί το ευρύτατο αυτό θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι σαφή τα ζητήματα, έχουν συστηθεί επαρκώς και αν συμφωνείτε Έχουμε δύο θέσεις σαφείς, είναι τη θέση του Συμβουλίου και η θέση της Κομισιόν. Και να το απλωστευσώ, πρέπει εμείς στην δική μας Επιτροπή να πάρουμε μια θέση. Γιατί καθώς υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ των δύο, θα περάσουμε σε ψηφοφορία για να δούμε τι μπορεί να σκεφτεί η Επιτροπή σε σχέση με τις δύο αυτές θέσεις. Δηλαδή, ποιοι είναι υπέρ της θέσης του Συμβουλίου ότι μπορούμε να έχουμε εκτελεστικέ πράξει ή να ποιοι είναι υπέρ τη θέση τη επιτροπή. Θα το ψηφίσουμε τώρα με ένα χειρός. Ποιο είναι υπέρ τη θέση του Συμβουλίου. Σηκώστε παρακαλώ τα χέρια γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Να μετρήσουμε favor de la, de la posición de la Comisión. Ποιο είναι υπέρ τη θέση τη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por tanto, por 8 votos. Μάλιστα. Οκτωψήφια έναντι τεσσάρων. Έτσι λοιπόν η εντολή που δίνεται στον διαπραγματευτή στην περίπτωση αυτή είναι να συνεχίσει στη γραμμή της Κομισιόν. Κάτι άλλο, μάλιστα. Είναι όλα σαφή, πολύ ωραία. Ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το οποίο είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχει. Θα σας πω εδώ. Σημείο 19. Ένα λεπτό, τελειώσαμε. Ανακοινώσει ε, για το τι θετήθηκε από τους ε, συντονιστές. Τα έχετε όλα αυτά. Κυρία Φράγα πρώτα εσείς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω μια διαμαρτυρία εδώ για την απάντηση που έστειλε ο Επίτροπος Ντεκούκτ στην επιστολή που στείλατε εσείς προηγουμένως ζητώντα την έκθεση αξιολόγηση για την Παππούα Νέα Γουινέα, έκθεση που είχε αναλάβει η ΓΑΜΑ Trade για να αξιολογήσει, συγγνώμη, λίγη ησυχία, για να αξιολογήσει την πιθανή δυνατότητα ή όχι της παρέκκλησης των κανόνων προέλευσης. Όλοι διαμαρτύρονται, αλλά όλοι μιλάνε. Λοιπόν, σα είχαμε ζητήσει να γράψετε μια επιστολή και να ζητήσετε αυτή την έκθεση. Ξέραμε ότι είχε ολοκληρωθεί και ο κύριος Δεκούκτ ε, πριν λίγες μέρες απάντησε και είπα ότι δεν μπορεί να στείλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίε με την Παππούα Νέα Γουινέα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό, γιατί οι διαπραγματεύσει με την Παππούα Νέα Γουινέα θα γίνουν στη συνέχεια. Αυτή είναι μια έκθεση που ε, έχει να κάνει με μια διαβούλευση και δεν εμπλέκει την Κομισιόν. Έτσι λοιπόν, ε, πραγματικά εγώ έχω ε, βαρεθεί λίγο αυτή τη στάση τη ΔΕΛΤΑ ΤΡΕΙΤ και του κ. Ντεγκούκτ και αυτή την έκθεση τον έχω εγώ μέσω τον ευρωπαϊκό κλάδο εδώ και ένα μήνα. Αλλά Έχω και ένα φίλο από την Αυστραλία, ερευνητή, που το έχει εδώ και ένα μήνα μέσω από τη παππούες Νέες Γουινέα. Και θέλω να πω ότι μου φαίνεται εξοργιστικό το πως η Κομισιόν και ο κύριο Ντεμπούκ συμπεριφέρεται σε αυτή την επιτροπή. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ορισμένου βουλευτέ. Έτσι λοιπόν, αυτή η μεταχείριση απέναντί μα δεν είναι σωστή. Γιατί έχω την έκθεση εδώ και ένα μήνα και ο κύριο Ντεμπούκ, επειδή ε, το ασκήθηκε πίεση, το έστειλε την περασμένη Παρασκευή και το έχουν όλοι οι Αυστραλοί από άλλε διόδε, και αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να το πετύχει, να το αποκτήσει την έκθεση αυτή. Θέλω να σημειωθεί στα πρακτικά και θέλω να πείτε στον κύριο Ντεκούκ ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχόμαστε αυτή τη μετεχείριση και θέλω επίση να είμαι ενημερώσει η Κομισιόν τι έχει γίνει με αυτή την έκθεση. Μάλιστα, κύριε Φράγκ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ε, ε, να ξέρετε τι έχει γίνει με αυτό. Να σας πω, όπως λέει και η κυρία Φράγκα, στείλαμε μία επιστολή στον Επίτροπο για να μας στείλει τις εργασίες και όπως είπε η κυρία Φράγκα, μας είπε όχι, δεν μπορεί να μας το στείλει την έκθεση αυτή, γιατί θα πρέπει πρώτερα να γίνουν συζητήσεις με την Παππούα Νέα Γουινέα και θα μας σταλούν αυτές οι πληροφορίες μέσω της ε, Επιτροπής Ίντα. Έτσι λοιπόν εμείς ε, στείλαμε μια επιστολή Λέγοντα ότι μας ε, φαίνεται παράδεκτη απάντηση γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η έκθεση ήδη έχει διανεμηθεί και πέρα από τον κλάδο το έχουν και άλλοι αυτό το έγγραφο. Έτσι λοιπόν ε, μας απαντούσε είναι ολόκληρο φιλμ, έτσι ολόκληρη ταινία. Και ε, μας απάντησαν ότι είναι, πρέπει να, να συναντηθούν με τη γραμματεία για να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι είναι απαράδεκτο, δεν έχουμε απολύτω τίποτα να συζητήσουμε για το πώ ε, αποκτήσαμε αυτή την έκθεση και ζητάμε επίσημα να παρουσιαστούν σε αυτή την Επιτροπή για να μας εξηγήσουν το όλο ζήτημα μας απαντούν και πάλι και μας λένε, και μάλιστα με κακό τρόπο μας απάντησαν, με άσχημο τρόπο, α, σιγά σιγά δεν ρυθμίζονται έτσι αυτά τα πράγματα, ηρεμήστε και την επόμενη μέρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να συναντηθούμε και μια μέρα να το συζητήσουμε αυτό με ηρεμία. Και πάλι μιλώ με τον Φιλίπ, συνομίλησα με τον Φιλίπ και είπαμε ότι δεν θα του απαντήσουμε σε αυτό και θα πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί του, απλώ να έρθουν εδώ στην Επιτροπή για να μα εξηγήσουν πώ έχουν τα πράγματα. Αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή. Η απάντηση σε αυτό το τελευταίο επιστολή μα ε, ήταν ε, η άμεση αποστολή του εγγράφου. Έτσι λοιπόν, ε, το βέβαιο είναι ότι αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώ απαράδεκτη. Το πώ συμπεριφέρθηκε ο Επίτροπο ε, σε αυτό το θέμα και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και συμφωνώ να στείλουμε μία επιστολή απευθεία στον κύριο Επίτροπο να εξηγούσουμε τι συνέβη και να του πούμε ότι απορρίπτουμε εντελώ αυτή τη διαδικασία. Συμφωνείτε. Not just the Commissioner, the the Commission, I think στο, στο, στον πρόεδρο της Επιτροπής ενδεχομένως. Στο... Ή να το στείλουμε στον ε, Επίτροπο με αντίγραφο στον πρόεδρο της Επιτροπής. For Για μένα είναι εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε να το στείλουμε κατευθείαν στον, ε, Πρόεδρο της Κομισιόν. entiendo, entiendo que lo que están sugiriendo es que una carta mía... Μία δική μου επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η κυρία Φραγκά εκτός μικροφώνου. <laughs> Κύριε Πρόεδρε, βλέπω στο, παρά, στο στα, στα πρακτικά το νέο χρονοδιάγραμμα για, για τη συνεδρία της Επιτροπής και βλέπω πάρα πολλές αλλαγές. Ε, είναι περίεργο αυτό, τόσες πολλές αλλαγές, γιατί συνέβη. Εντάξει, το συζητήσαμε και με τους συντονιστέ σήμερα το πρωί. Οι αλλαγέ έγιναν ε, λόγω της συμφωνίας ε, των Προέδρων, της διάσκεψης των Προέδρων συμφωνήθηκαν εκείνα κριτήρια σε σχέση με τι ημέρε συνεδρίαση των επιτροπών. Θα είναι Δευτέρε και τρίτε, ή Τετάρτε και πέμπτε, αλλά δεν θα συνδυάζονται ημέρε. και βάσει αυτών από τον Απρίλιο γίνονται αυτέ οι τροποποίησει. Επιβλήθηκαν και το είπαμε σήμερα το πρωί αυτό στους ότι για φέτο δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, αλλά για το επόμενο έτος θα προσπαθήσουμε οι ημέρε να βολεύουν εμά και όχι άλλου. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συνεδριάσουμε στις 20 Μαρτίου το απόγευμα και στις 21 το πρωί και το απόγευμα. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που μας αντέξατε και ευχαριστεί ο Πρόεδρος και τους ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.